So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this morning's meeting. Our first item on the agenda, point 13, is the annual report on competition policy, which is an important annual report which comes before our committee and obviously then on... Καλημέρα σας. Η σημερινή συζήτηση είναι η δεύτερη συζήτηση από τους συναδέλφους και από ό,τι κατάλαβα έχει διοργανωθεί, έχει προβλεφθεί μάλλον συνεδρίαση ανάμεσα στους κοιόδης γιατί έχουν κατατεθεί 221 τροπολογίες. Να ρωτήσω λοιπόν τον εισηγητή, τον κύριο Ρημό να λάβει το λόγο. Um, Στα γερμανικά θα μιλήσω. Αυτή η έκθεση ήταν ε, πολύ θετική γιατί όλα έγιναν επικοδομητικά και με τους σκιώδεις και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Οπότε πάμε για καλή έκθεση. Αφενός διότι διαπαραταξιακά θεωρούμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι, είναι λειτουργική και η Κομισιόν συμβάλλει πολύ σημαντικά σε αυτό. Έχει λοιπόν θεμελιωδώς καλά στοιχεία. Πιο πολύ εστιάσαμε στο μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού αυτό έδειξαν συζητήσεις και περισσότερες τροπολογίες. Το κεντρικό θέμα είναι ότι και θα το συζητήσουμε σε βάθος στην επόμενη συνάντηση των σκιωδών και θα μας πούν και οι σκιώδες απόψε είναι ο ψηφιακός τομέας της ε, πολιτικής ανταγωνισμού όπου έχουμε προκλήσεις που δεν γνωρίζουμε στην κλασική πολιτική συγχώνευση του WhatsApp και του Facebook, παράδειγμα. Δύο μεγάλες επιχειρήσεις που τώρα συγχωνεύονται σε μία ακόμα μεγαλύτερη επιχείρηση. Η μία δίνει υπηρεσίες δωρεάν. Το Messenger Dienst και με το κλασικό δίκαιο του ανταγωνισμού που πρόκειται για μερίδια αγοράς κλπ. Ε, δεν αντιμετωπίζεται, δεν έχουν τζίρο δηλαδή. Οπότε το δίκαιο ανταγωνισμού όπως ίσχυε μέχρι τώρα δεν μπορεί να τους καλύψει. Ε, δεν μπορεί να λάβει υπόψη την επίδραση που έχουν όλα αυτά στους καταναλωτές και τους χρήστες. Σε αυτό το τομέα θα συζητήσουμε πολλές συγκεκριμένες υποθέσεις ε, όπως οι πλατφόρμες ε, και πώς λειτουργούν για τη στέγαση και τον τουρισμό και πώς θα πρέπει η πολιτική ανταγωνισμού να αντιμετωπίσει τη δημιουργία των δικτύων, την κάλυψη της υπαίθρου προς το δημόσιο συμφέρον και πότε παρεμβαίνει το δίκαιο ανταγωνισμού και πότε είναι στο προσκήνιο η λειτουργία της αγοράς. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο διαπραγματευτικό ζήτημα και ε, ξαναγυρίζω σε μια βασική συζήτηση που έγινε για την έκθεση αυτή. Ένα θέμα που συζητούμε είναι το εξής. Το δίκαιο ανταγωνισμού που λειτουργεί τόσο καλά μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον ε, με ευρύτερη βάση όπου θα προσέχουμε και περισσότερο θέματα κοινωνικά, τις κοινωνικές πλατφόρμες που αποκτούν μεγαλύτερη πολιτική σημασία ε, ναι, τα πολιτική προπαγάνδα, ε, τα θέματα του Brexit, όπως είναι ένα παράδειγμα που αντιμετωπίστηκε από το, τις πλατφόρμες αυτές. Και γενικά το δίκαιο ανταγωνισμού είναι το σωστό πλαίσιο ή αν διευρυνθεί περισσότερο για να συμπεριλάβει περισσότερα θέματα αυτό θα είναι κακό Θα μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή ένα δικαίωτο ανταγωνισμού που να προστατεύει και τη δημοκρατία. Πολλά ε, θέματα άπτονται ε, εδώ. Έχουμε και στον τομέα της γεωργίας ε, θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Τα τελευταία 30 χρόνια το μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής σπόρων ανέβηκε στο 62% της ε, παγκόσμιας αγοράς ε, σπόρων και έτσι μειώνεται και η ποσότητα και το είδος των σπόρων. Αυτό δεν είναι καθαρά οικονομικό θέμα με ποσοστό τζίρου, μερίδια αγοράς κλπ. Πρέπει να δούμε και άλλα θέματα, δηλαδή αυτές οι συγκεντρώσεις θα πρέπει ίσως να κρίνονται με άλλα κριτήρια και να δούμε και ποιο είναι το σωστό πλαίσιο για να κρίνονται. Ε, διότι βέβαια ε, θα πρέπει να μην γίνει πολύ συγκεχημένο ε, από την πολίτη διεύρυνση το δίκαιο ανταγωνισμού. Θα πρέπει να βρεθεί δηλαδή μια σωστή ισορροπία. Πάντως οι συζητήσει μέχρι τώρα ήταν πολύ επικοδομητικές, ξαναλέω. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρεμάν. Για το ΕΛΚΑ, Σκιώδης, ο κύριος Χάκμα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για αυτήν την έκθεση που προετοίμασε, αλλά και για την συζήτηση που έχει ξεκινήσει. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να συμβάλλουμε όσον αφορά, σημαντικά, ε, όσον αφορά αυτή τη σημαντική ε, έκθεση. Κάποιες σκέψεις από τη δικιά μου πλευρά όμως. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της Κομισιόν όσον αφορά την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Εμείς είμαστε αυτοί που κρίνουμε ας πούμε τι κάνει η Κομισιόν. Να μην λέμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερος εκείνο ή το άλλο. Και δεν χρειάζεται να πολιτικοποιήσουμε βέβαια τις αρχές του ανταγωνισμού. Όταν ε, ε, υπεραμεινόμεθα της ανεξαρτησίας της Κομισιόν ε, σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού, στην ουσία κάνουμε καλό στην πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, αλλά ίσως ακόμα καλύτερα είναι να εξασφαλίσουμε νέες εισόδους στην οικονομία και μάλιστα να διασφαλίσουμε τη διασυνοριακή ανάπτυξη της οικονομίας. και ενταγμένο στην πολιτική ανταγωνισμού στην ουσία είναι το πλήρες φάσμα της οικονομίας. Και όταν ε, κάνουμε νέα βήματα, ας πούμε, όσον αφορά την ενέργεια και την αγορά ενέργειας, ε, είναι κάτι σοβαρό. Και ε, βεβαίως και η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη αυτή την ενεργειακή αγορά υπό το πρίσμα της διακυβέρνησης. Εμείς ε, θέλουμε δραστηριότητα σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το πεδίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, στις τροπολογίες μας λέμε ότι δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές θεωρήσεις ε, αλλά να ληφθούν υπόψη τα αντικειμενικά ε, ε, στοιχεία. Είμαστε υπεύθυνοι και για το κλίμα και για την ενέργεια ε, και για τα κοινωνικά στοιχεία που πρέπει να αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει, να αναλάβει δράση σε, αυτές τις, σε αυτά τα πεδία. Επίσης υπογραμμίζουμε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να δράσουμε κατά των κυβερνήσεων που ακολουθούν φορολογικές πολιτικές που στόχο έχουν την στερεύλωση του ανταγωνισμού και ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν μονάχα και είναι ε, ε, ευθύνη μόνο των κρατών και επομένως δεν θα πρέπει είτε το Κοινοβούλιο είτε η Κομισιόν να ανακατευτούν σε αυτά. Ε, η σκέψη μας είναι ότι θα πρέπει αφενός να κατοχυρώσουμε τον σεβασμό της ανεξαρτησίας της ε, Κομισιόν ε, και από την άλλη ε, να παραδεχτούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ένα δυναμικό στοιχείο της οικονομίας, να διευκολύνουμε νέες εισόδους ε, στα πλαίσια βέβαια αυτών που αναφέρατε και εσείς για την ψηφιακή οικονομία και για τις ψηφιακές πλατφόρμες και για τις ενεργειακές αγορές. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε σαφείς και να βοηθήσουμε, να καθοδηγήσουμε την Κομισιόν για, την, για τον σωστό ανταγωνισμό, τον καλό, μεγάλο ανταγωνισμό, ο οποίος είναι καλός για την οικονομία. Thank you, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάκμαρ, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη συζήτηση, εδώ πρόκειται για ε, έκθεση η οποία είναι περιβαλλοντικά φιλική ε, και επομένως δεν έχουμε ιδιαίτερους προβληματισμούς Βεβαίως εμείς ως σοσιαλιστές ε, εστιάζουμε σε τροπολογίες οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένα πεδία που είναι σημαντικά και για την ομάδα μας αλλά και για τους πολίτες. το θέμα της ε, φορολογίας ας πούμε είναι σημαντικό. Ναι, βεβαίως μπορεί να είναι εθνική ε, ε, αρμοδιότητα, αλλά μπορεί να έχει και αντίκτυπο σε συνολικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φορολογία ως στοιχείο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Επίσης το θέμα της ψηφιοποίησης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. και δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, το θέμα των υφιστάμενων ε, κρατικών επιχορηγήσεων. Αυτό ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μην αμαυρώνει την, ή να μην αλλοιώνει μάλλον την εικόνα. Τέλος. θα θέλαμε να ε, είναι πιο ξεκαθαρισμένος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αναφέρεται δηλαδή πιο σαφώς η ε, δύναμη συναπόφασης που έχει το Κοινοβούλιο. τα στοιχεία τα οποία αφορούν ε, το πλαίσιο του ανταγωνισμού δεν είναι εκτός πεδίου γιατί ε, στόχο έχουν να διευκολύνουν τους πολίτες, να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Εμείς είμαστε ε, σοσιαλιστές και αυτό μας ενδιαφέρει. Και ευελπιστούμε λοιπόν ότι στις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών ε, θα γίνουν πιο ξεκάθαρες και οι θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και οπωσδήποτε ότι θα προσεγγίσουμε οι μεν τους δε. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καλύψουμε το συμφέρον των πολιτών. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχουν και πολιτικές προτεραιότητες ε, όπως είναι, που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό όπως είναι ε, η ενίσχυση της ε, καινοτομίας, είναι η εσωτερική αγορά και κυρίως η επαναδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το ECR έχουμε κάποιον εδώ. Όχι. Άλντε υπάρχει κάποιος. Όχι. Γκουε. Η κυρία Λόπες Περμίγιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρεμόν τον εισηγητή για την ε, εργασία του. Ναι, πρόκειται για ένα πολύ ε, περίπλοκο ζήτημα, ε, δύσκολο στην διαχείρισή του και την αντιμετώπιση του γιατί εδώ εκδηλώνονται διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το φάσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το μέχρι που ε, θα πρέπει να φτάνουν αυτές οι πολιτικές τουλάχιστον νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, και στις ευχαριστίες ε, προς την αρμόδια Επίτροπο και για τη θέση της και για τις σχέσεις που έχει με την Επιτροπή μας. Ωστόσο, Πιστεύω ότι δυστυχώς οι συμφωνίες, οι υπόλοιπες δηλαδή συμφωνίες οι οποίες υλοποιούνται εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι δύσκολο να επιτευχθούν κυρίως γιατί τα σημεία εκκίνησης σχετικά δηλαδή με το τι είναι η πολιτική ανταγωνισμού ε, δυσκολεύουν την ε, πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να αναφερθώ σε δύο στοιχεία όσον αφορά ε, την ε, πολιτική ανταγωνισμού ε, εν γέννη. Πρώτον, η πολυμορφία, η ποικιλομορφία και όσον αφορά τη μορφή και όσον αφορά τον ορισμό. Ο ορισμός πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι σταθερό. Δεν μπορεί να δουλέψουμε σαν να ήταν μια συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία δεν αλλάζει. Δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι επιμένουμε πολύ υπερβολικά ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι κάτι τεχνικό. Εγώ όμως λέω ότι αναμφίβολα οπωσδήποτε η πολιτική ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα πολιτικό θέμα γιατί και έχει αποτελέσει ε, το, το επίκεντρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι δυνατόν να ε, την απογυμνώσουμε από τις αρχές της και να την απομακρύνουμε από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ε, λόγο όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και όσον αφορά τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση που θα πάρει η πολιτική ανταγωνισμού. Ε, πιστεύουμε ότι ναι, αυτή η πολιτική θα πρέπει να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, την πλειοψηφία και θα πρέπει να αγωνιστεί κατά ε, των αυξήσεων τιμών ε, ενέργειας που καταδικάζουν ε, στην ενεργειακή φτώχεια, να αγωνιστεί κατά της καταχρηστικής αύξησης τιμών έτσι ώστε γενικότερα οι πολίτες, γενικότερα οι γεωργοί να μπορέσουν οπωσδήποτε να έχουν τα θετικά, το θετικό θετικό αντίκτυπο μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού. Επίση, θα πρέπει να μειώσει την διάσταση, ψηφιακή διάσταση, την ε, ψηφιακή ε, ε, διαφορά που υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν θα ε, αποτελέσει ε, ακόμα μία μπάλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο τώρα που πλησιάζουμε και στα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Θα πρέπει ε, η παρέμβαση στην πολιτική διαδικασία να είναι ουσιαστική. Να υπενθυμίσω ότι η αρχή της πολιτικής ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή. Να παρεμβαίνει στις αστοχίες της αγοράς έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα καλό πλαίσιο για την αγορά και για τους καταναλωτές, δηλαδή για τους πολίτες. Κατά την έννοια αυτή θα αγωνιστούμε και ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν ε, ευρείες συνενέσεις και θα είμαστε πάντα στη διάθεση του εισηγητού για να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον εδώ από το ENF. όχι. Κανείς. Ωραία, λοιπόν, ας περάσουμε στο Catch the Eye. Εξ ονόματος του, κυρί... του ΕΛΚ, ο κύριος Βάμπ θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καταρχάς συγχαρητήρια στον εισηγητή και στους εσκιώδεις. Πιστεύω πως η έκθεση και οι τροπολογίε είναι πολύ καλές ε, και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θέλω να εστιάσω σε ένα σύνολο βασικών τροπολογιών που θεωρώ πως είναι σημαντικές. Η μία είναι το ένα σύνολο είναι ότι ε, έχουμε το 30, την 37 ε, και λοιπές ε, εστιάζει στο τι ακριβώς είναι η, πολιτική ανταγωνισμού εστιάζει περισσότερο στον κλασική ορισμό δεν πρόκειται για κοινωνικά δικαιώματα ή για τίποτα άλλο αλλά για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι αγορές υπό κανονικές συνθήκες και αυτό είναι και το καλύτερο για όλους μας για το περιβάλλον, για τους πολίτες και τους καταναλωτές. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε αυτό το σύνολο τροπολογιών. Το δεύτερο, ε, ήδη το ανέφερε ο Μίχελ Ράιμον και άλλοι συνάδελφοι, ότι δηλαδή προσπαθούμε να προλάβουμε την ψηφιακή ε, καινοτομία, να δούμε απαντήσεις σε περίπλοκα ζητήματα και θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία να μην προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε όλα ταυτόχρονα, αλλά ούτε και να μην προσπαθήσουμε ή να διστάζουμε υπερβολικά να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η πρόταση της Κομισιόν είναι καλός ε, τρόπος να προχωρήσουμε, είναι κάπως διστακτικό, ε, διστακτική προσπάθεια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και υπερβολικά. 54, 64 και 86 τροπολογίες δείχνουν ότι χρειαζόμαστε μία ε, επιφυλακτικότητα όταν προσεγγίζουμε νέους τομείς και ίσως να είναι αυτό απαραίτητο όταν πλησιάζουμε, ασχολούμαστε μάλλον με τον τομέα του ε, ηλεκτρονικού εμπορίου και του τομείς της, ε, το θέμα μάλλον του ανταγωνισμού. Θα ήθελα να εστιάσω στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είδαμε για την οδηγία περί ζημιών κοντεύουμε πια να φτάσουμε στο τέλος, αλλά τα κάτι μέλη προκαλούν ε, καθυστερήσεις και δεν θα είμαστε τόσο αποτελεσματικοί εάν ε, καθυστερήσουμε υπερβολικά στην εφαρμογή. Τέλος, να στηρίξω και τον ε, σκιώδη μας τον κύριο Χόκμαρ που έκανε εξαιρετική δουλειά με τις τροπολογίες του για τη στρατηγική για τις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε θέματα ανταγωνισμού εάν προχωρήσουμε ταυτόχρονα, μάλλον γρηγορότερα, σε κάλυψη ε, Wi-Fi πέμπτης γενεάς. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν εδώ. Τελευταίο μου σημείο προς τον εισηγητή και τους σκιώδεις και ίσως και προς την Κομισιόν ότι πιστεύουμε πως στον τομέα της ε, ε, πολιτικής ανταγωνισμού της παραδοσιακής ε, των καρτέλ έχουμε αυξανόμενο αριθμό καρτέλ. Μια ερώτηση είναι, υπάρχουν λιγότερα καρτέλ ή υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες για, τα κράτη, για τις αρχές ανταγωνισμού να ανακαλύψουν την ύπαρξη αυτού του καρτέλ. Γιατί είναι εύκολο να λέμε ναι, ναι η οικονομία είναι, δεν πάει καλά, υπάρχουν περισσότερα καρτέλ αλλά ε, δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Εν πάση περιπτώσει να γίνεται μια... Ε, μια αξιολόγηση της κατάστασης από καιρού εις καιρών για να βλέπουμε τι συμβαίνει με τα καρτέλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Αλλιώς να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Το θέμα είναι πως ε, η πολιτική ανταγωνισμού βρίσκεται στην καρδιά της υπεράσπιση της ευνοίας αγορά. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ε, ε, δυσλειτουργούσα ε, ενιαία αγορά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και την πολιτική ανταγωνισμού για να μπορούμε αυτό να το υλοποιήσουμε. Και γι' αυτό και συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή ότι πρέπει να μπορούμε να ανοιχνεύουμε τα καρτέλ και τις προτιμησιακές αντιμετωπίσεις για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Αλλά στην σημερινή αγορά είναι δύσκολο κανείς να πει τι είναι καρτέλ και τι δεν είναι. Ο πολιτική ανταγωνισμού αφορά δε και την ενθάρρυνση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, αρμοδίων αρχών εν περιπτώσει, να είναι πιο δραστήριες στα ίδια τους τα κράτη-μέλη και άρα να προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών κανόνων ανακράτως μέλος για να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα εφαρμόζεται με τρόπο που να είναι ξεκάθαρος για όλους. Και νομίζω πως το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για τη, και, και οι ελάχιστες νομικές προδιαγραφές είναι ευπρόσδεκτες ε, για να μπορέσουμε να ε, τις ε, τοπικές μάλλον τις ανακράτους αρχές αρμόδιες για τον ανταγωνισμό να δράσουν περισσότερο. Τέλος, θα πρέπει η Κομισιόν να βλέπει τις υποθέσεις που έχουν συστημικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά. Σε κάθε υπόθεση θα πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και το τέλος. Και γι' αυτό είναι σημαντικό στην επιλογή των υποθέσεων να υπάρχει τελικά ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να το δει. Ε, Είναι σημαντικό λοιπόν τα κράτη-μέλη να μπορούν να βλέπουν, μάλλον και ο κόσμος να μπορεί να βλέπει ποια είναι η εξέλιξη τελικά και να γίνεται αυτό έγκαιρα και με τρόπο που να έχει συστημική σημασία και επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας το αυτό, αν πάρουμε την τωρινή μη αυθαίρετη προσέγγιση ε, δεν το καταφέρνουμε πάντοτε αυτό. Ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν πριν επανέλθουμε στον εισηγητή μας. Εξ ονόματος στην DG Comp, ο κύριος Λίντιμπεργκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και όλη και την Επιτροπή διότι έκανε ευρεία και σε βάθος ανταλλαγή ε, απόψεων για αυτό το θέμα και όλα τα άλλα. Η Κομισιόν αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτή την ανταλλαγή που είναι σημαντικός παράγων και για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και την Κομισιόν γενικότερα για να ελέγχει την επιβολή των πολιτικών της ε, πάνω στην πραγματικότητα και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Χαιρόμεθα διότι φαίνεται να υπάρχει ευρεία συνένεση για τα σημαντικά θέματα που είναι στο προσκήνιο της έκθεσης και ε, βέβαια υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα που συμπεριελήφθησαν και στη σημερινή συζήτηση και στις τροπολογίες. Να αναφέρω γρήγορα ορισμένα θέματα χωρίς να είναι εξαντλητική η παράθεση. Η Κομισιόν θεωρεί ότι έγινε μια γόνιμη συζήτηση για τα όρια δικαιοδοσίας της πολιτικής ανταγωνισμού. Η Κομισιόν δεν πιστεύει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να περιορίζεται στην στενή εξέταση μόνο τιμών παραγωγής Παράμετροι όπως επιλογή, καινοτομία, ποιότητα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτές οι παράμετροι επιτρέπουν να ληφθείουν υπόψη στρεβλώσεις της αγοράς που με τη σειρά τους επηρεάζουν θέματα όπως το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία. Αυτό υπογραμμίζεται και από την εξέταση από την Κομισιόν μεγάλων συγχωνεύσεων Bayer Μουντσάντο, Ντάνι και China Σιντζίντα όπου η Κομισιόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο κόστος για τους αγρότες, αλλά και για τις δυνατότητες των ε, γεωργών να επιλέγουν. Συμφωνούμε όλοι ότι η ψηφιοποίηση θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις για να γίνουν κατανοητά όλα τα σχετικά στοιχεία και να υπάρξουν και έγκαιρα συμπεράσματα που θα επηρεάσουν την αγορά. Αυτή είναι συνεχιζόμενη εργασία. Γιατί έχουμε πολύ σύνθετες περιπτώσεις. Ανέφερα για παράδειγμα την έρευνα για την Google έρευνες ε, που δεν γίνονται τώρα πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, δεν είναι ένα έργο που θεωρείται ολοκληρωμένο και γι' αυτό η Επίτροπος Βέσταγκερ ε, κάλεσε τρεις εμπειρογνώμονες για να ε, κάνουν περαιτέρω ανάλυση των προκλήσεων του ψηφιακού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Και γι' αυτό μεταξύ άλλων η Επίτροπος Βεστάγκερ θα συγκαλέσει τον Ιανουάριο μια διάσκεψη όπου θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα αυτά περισσότερο. Ε, σίγουρα υπάρχει και θέμα ταχύτητας και έγκαιρης ολοκλήρωσης των ερευνών και βλέποντας και τι τροπολογίες, ε, τονίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κομισιόν, η οποία εξετάζει όλες τις δυνατότητες ε, για να επιταχύνει την ταχύτητα των ερευνών. Ε, από την πρόσβαση στο φάκελο μέχρι διαδικασίες συνεργασίας και περαιτέρω εξέταση των ενδιάμεσων μέτρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και οι πιο γρήγορες περιπτώσεις ε, δεν πρέπει να ε, περιορίζουν την ποιότητα. Όλα τα σχετικά στοιχεία μιας υπόθεσης θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, συνολικά. Για τα καρτέλ θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός είναι ένας τομέας προτεραιότητας, πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι για την Κομισιόν προτεραιότητα. Είναι πηγή ανησυχία ε, τρόπον την αν μετά από 10 και παραπάνω χρόνια έντονη επιβολή των κανόνων η κατάσταση στα καρτέλ θα ήταν ακριβώ η ίδια όπως και πριν από την αρχή της δεκαετίας τη επιβολή των νέων μέτρων. Η αποτροπή επίσης πρέπει να έχει αντίκτυπο. Τώρα δεν είναι πιθανό ακόμα και η ισχυρότερη επιτροπή, αποτροπή να ε, καταρρύψει όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια ε, στα, για, στη δημιουργία καρτέλ. Γι' αυτό η Κομισιόν τώρα θέλει να ε, ε, εστιάσει τις παρεμβάσεις, δηλαδή μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μέχρι εξέταση των προγραμμάτων συγκέντρωσης και ε, σίγουρα και τα μέσα και οι μηχανισμοί ανταγωνισμού θα είναι πολύ σημαντικοί. Ο προσανατολισμός στην ενιαία αγορά μέσα από τις διάφορες ε, παραμέτρους της επηρεάζει την πολιτική ανταγωνισμού. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και πάλι για τη μεγάλη υποστήριξη που δόθηκε στην οδηγία Ίσιαν Συν ε, που βοήθησε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές ε, αρχές ανταγωνισμού και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα μέτρα θα εφαρμόζονται. Η Κομισιόν θα συνεργαστεί και στο μέλλον και με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις τις επόμενες εβδομάδες για την οριστικοποίηση της έκθεσης. Και άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την προθυμία σας ε, για διάλογο. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Άλλον δεν βλέπω να ζητεί το λόγο. Ο κύριος Ραϊμόν θα κλείσει τη συζήτηση. Ο, α, ο, ο, ε, ε, νομίζω ότι ε, μπορούμε να κάνουμε μια ιδεολογική συζήτηση για όλο το θέμα, το, το θέμα. Μας ενδιαφέρει μας ενδιαφέρει πολύ ε, να μην είμαστε φονταμενταλιστές όσον αφορά ε, την αντιμετώπιση του θέματος. Ο κύριος Φάμπ λέει ότι ε, μέσω της τροπολογίας του ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και εξωτερικά στοιχεία στην πολιτική ανταγωνισμού. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι λοιπόν να προχωρήσουμε και να ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρημόν. Η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ για την έκθεση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια θα περάσει μάλλον τον Ιανουάριο του 2019. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Σας ζητώ πάντως ε, να παραμείνετε στην αίθουσα γιατί το επόμενο θέμα ε, είναι, ε, προβλέπει την παρουσία του Προέδρου του Eurogroup στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου και αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 10 ακριβώς. Ευχαριστώ.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 Συνάδελφοι, να καλωσορίσω θερμά σήμερα εδώ τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένα, που είναι εδώ για τον τακτικό οικονομικό διάλογο. Όπως γνωρίζετε έχουμε, διετή, έχουμε ε, ετήσιο οικονομικό διάλογο με το Eurogroup που γίνεται στις αρχές και στο φθινόπωρο κάθε χρόνο. 21 Φεβρουαρίου ήταν η προηγούμενη μας συνάντηση. Ε, σημαντικό σήμερα είναι να μιλήσουμε για τα θέματα για το εξάμεινο, για τους συστάσεις αναχώρα, για τον προϋπολογισμό και αλλά και για να κάνουμε μια έναν ε, απολογισμό πριν από την διάσκεψη κορυφής ε, στο, του Δεκεμβρίου να μιλήσουμε για την ταχύτητα εφαρμογής του ε, πλαισίου εποπτείας στην Ελλάδα. Από ό,τι κατάλαβα χτες είχατε σημαντική συζήτηση για το backstop, το προστατευτικό ε, καθεστώς, καθώς και για τη μεταρρύθμιση του ESM και την ε, ιδέα της δημοσιονομικής δυνατότητας. Κάνουμε εξαιρετικά ε, προσπάθειες για να επιταχύνουμε την δέσμη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου και έχοντας όλα αυτά υπόψη, σήμερα θα πρέπει να συμβάλλουμε στη μεταρρύθμιση της ε, ΟΝΕ. Ναι. Πολύ μας ενδιαφέρουν τόσο, όσα θα μα πείτε, γιατί ελπίζουμε ότι η προσπάθεια που εμείς καταβάλουμε θα συνοδευτεί από κάποια βήματα μπροστά στη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ. Ναι. Φυσικά το προστατευτικό καθεστώ είναι το backstop, είναι σημαντικό στοιχείο. Η ε, πρόορη εφαρμογή αυτού ε, κατά ένα-δύο χρόνια ε, θα είναι κάτι το θετικό. Εν πάση περιπτώσει είμαστε μέσα ε, ε, στην μεταρρύθμιση της ε, ΟΝΕ. Ναι, υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία. Να πω μόνο δύο λόγια. Όταν διάβασα τις χριστιανέ σας παρατηρήσεις, Βεβαίω μα ενδιαφέρει πολύ και θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της Κομισιόν για το, και του ESM. Η διατήρηση βεβαίως των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και ελπίζουμε πως αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα καταλήξουν στο να μειώσουν το ρόλο τη που ήταν πολύ σημαντικός πρόσφατα. Αν θυμάμαι καλά το ρόλο που έχει παίξει η Κομισιόν στη διάρκεια του τελευταίου προγράμματος για την Ελλάδα με τον κύριο Κοστέλο, ε, δεν θα κατεβούμε από αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε ότι θα το υπερβούμε. Θα μας πείτε λοιπόν κάποια πράγματα, καθώς και τα διάφορα στοιχεία της συζήτηση που κάνατε. καθώς και τη γνώμη του Eurogroup σε αυτή τη δημοσιονομική φάση, γιατί ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε περίπλοκα και ελβέστητα θέματα. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Ρομπέρτο. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στην Επιτροπή ε, ΕΚΟΝ για τον διετή, δι, ε, μάλλον τον ε, ετήσιό μας διπλό διάλογο. Έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία και τα βασικά στοιχεία επί των οποίων εργάζεται το Eurogroup. Η Ευρωζώνη επεκτείνει την ανάπτυξή της. Η οικονομία αναπτύσσεται για 22 διαδοχικά τρίμηνα έχουμε βασικές θετικές σχέσεις και αυτό σημαίνει ε, κάποια κανονικότητα σε σχέση με την ισχυρή απόδοση του 17 όταν η ανάπτυξη έφτασε σε ανώτατο επίπεδο για 10 χρόνια. Επίσης είναι θερδικό που βλέπουμε το αμαδοποιημένο ΑΕΠ να αυξάνεται. Επίσης οι οικονομίες μας δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, τα μυρωμίστια αυξάνονται και υπάρχουμε ε, και αυτό μάλλον ευνοεί το ε, διαθέσιμο εισόδημα. Οι επενδύσεις επίσης ε, επεκτείνονται και οι προβλέψεις δείχνουν μια βιώσιμη θετική ε, προοπτική παρά ενδεχόμενους εξωτερικούς ε, παράγοντες κινδύνου. Συμφωνώ με αυτή την αξιολόγηση. Οι οικονομίες μας ε, παραμένουν σε μια θετική ε, πορεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε και θα πρέπει να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές, να μην επαναλάβουμε σφάλματα του παρελθόντος και να μπούμε και να προωθήσουμε υπερκυκλικές πολιτικές θα πρέπει οι αυτόματοι σταθεροποιητέ μα να μπορούν να λειτουργήσουν σε περιπτώσει κρίση χωρί να αμφισβητείται η βιωσιμότητα τη ε, ε, οικονομία. Επίση, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικέ μα θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη. Αυτό θα απαιτήσει κάποιε προσπάθειε, λαμβάνοντα υπόψη ε, ότι υπάρχουν κάποια ε, ε, μικρά προβλήματα. Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι χώρες ε, και τα κράτη-μέλη τα οποία υπερβαίνουν τα δημοσιονομικούς τους μεσοπρόθεσμους στόχους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικό χώρο για να δημιουργήσουν, μάλλον να καλύψουν τα κενά των επενδύσεων. Γι' αυτό υπάρχει και κοινή δημοσιονομική πολιτική και σχετική κανόνες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ανισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση είναι ε, διφυής. Δηλαδή η σύγκληση ε, πρέπει να ισχύει και για τις πλεονασματικές χώρες και για τις ελληματικές χώρες. Στο Eurogroup έχουμε εστιάσει στο σχέδιο προϋπολογισμού των χωρών και βέβαια αναπόφευκτα εστιάσαμε στο δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ιταλίας. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα δεν βελτιώνει την κατάσταση σε σχέση με την χρηματοδότηση και το βλέπουμε αυτό στις αγορές καθημερινά. Αυτό σημαίνει σημαίνει πως δεν έχουν αυληθεί οι ανησυχίες σε σχέση με την δημοσιονομική στρατηγική της Ιταλίας. Τώρα περιμένουμε την γνώμη της Κομισιόν για το αναφερειμένο σχέδιο της Ιταλίας, το οποίο αναμένεται αύριο μαζί με τις απόψεις ε, για τις γνωμοδοτήσεις μάλλον για τα σχέδια προπολογισμού των άλλων χωρών. Θα τα συζητήσουμε το Δεκέμβριο. Ε, ακατανοώ και μοιράζομαι τις ανησυχίες της Ιταλίας για την ε, μικρή ανάπτυξη και τα περίπλοκα κοινωνικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ε, διακινδυνεύσουν την πορεία της δημοσιονομικής εξυγίασης. Οι κανόνες είναι ένας, ένα μέσο για την επίτευξη ενός στόχου. Θέλουμε οικονομική ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η προσχόληση σε αυτούς δεν είναι ε, συμφέρον κάθε χώρας χωριστά. Είναι συνολικό συμφέρον όλων μας. Η κρίση μας δίδαξε ότι σε νομισματική ένωση είναι σημαντικό να ασκούμε υπεύθυνη πολιτική η οποία δεν σταματά στα σύνορα της χώρας μας. Αυτό το μάθημα το έχουμε μάθει πολύ καλά και πολλές χώρες έχουν επιβάλει και εφαρμόσει οδυνηρέ αλλά απαραίτητε μεταρρυθμίσει μετά από την κρίση. Να πω τώρα δύο λόγια για την Ελλάδα. Τον Αύγουστο φέτο η Ελλάδα επιτυχώ ολοκλήρωσε το οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογή που ήταν το τελευταίο πρόγραμμα ε, τέτοιο πρόγραμμα που λειτουργούσε στην ε, Ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν πέρασε εύκολες μέρες και οι Έλληνες πολίτες ακόμη λιγότερο, γιατί η χώρα χρειάστηκε να ε, διανύσει μια πορεία μεταρρύθμισης. Όμως τώρα φαίνεται τα πράγματα να είναι θετικά, η ανάπτυξη έχει επιστρέψει υπάρχουν ε, θετικές εξελίξεις, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, καθώς και το πλεόνασμα 3,5% έχει επιτευχθεί. Τον Ιούνιο το Eurogroup αποφάσισε διάφορα στοιχεία που σφράγισαν την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Αυτό σήμαινε και την τελευταία ε, ε, δόση που κάλυπτε τις ε, δημοσιονομικές ανάγκες για 22 μήνες. Ε, περιελάμβανε και τα μέτρα ώστε η Ελλάδα να μπορεί να ε, είναι βιώσιμη για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν την, ε, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σε αυτή την πορεία να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτές τις δημοσιονομικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστούν οι προοπτικές των πολιτών ε, ε μακροπρόθεσμα. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα. Η, προ... η πρόοδος της Ελλάδας θα αξιολογιστεί υπό την Εθνική Διαδικασία Εποπτείας και περιμένουμε αύριο την πρώτη σχετική έκθεση. Το Eurogroup θα εκτιμήσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα επί τη βάση των εκθέσεων που έχει προετοιμάσει η Κομισιόν ε, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμούς. Και τώρα να πω δύο λόγια για τις διαρθρωτικές πολιτικές. Οι υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές είναι απαραίτητες, αλλά όχι επαρκείς για να εξασφαλίσουμε τη στεναρότητα και την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας. Ε, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνοδεύονται από φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται πολιτικές που να προωθούν την παραγωγικότητα και άρα την ε, σημαντική ανάπτυξη. Να, να, να βελτιωθούν να βελτιωθεί το θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, να αρθούν οι φραγμοί και τα εμπόδια στι και, στην, και να, επίσης να προωθήσουμε την καινοτομία. Για αυτό το λόγο το Eurogroup κάνει τακτικές θεματικέ συζητήσει με τη συμμετοχή ε, καθηγητών και ειδημόνων. Είναι εξαιρετική ευκαιρία για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να ακούσουμε απόψει και συμβουλέ από εξωτερικούς εμπειρογνώμονε. Και τώρα θα στραφώ στην κατάσταση της συζήτησή μας για την ευάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Μια ανθεκτική Οικονομική και Νομισματική Ένωση απαιτεί ε, υγιείς οικονομικές πολιτικές. Από τον Ιούνιο φέτος το Eurogroup έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια σε αυτό. Ή, ε, περιμένουν, περιμένει ο, οι, οι ηγέτες συγκεκριμένα αποτελέσματα για το Δεκέμβριο. Ε, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του προστατευτικού καθεστώτος για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Ε, ε, το Eurogroup συζητά τις τελευταίες λεπτομέρειες αυτού του προστατευτικού καθεστώτος. Θα έχουμε μια πιστοτική γραμμή από ό,τι φαίνεται το μέγεθος της οποίας θα καθορίζεται από το ενιαίο Ταμείο θα χρειάζονται συγκεκριμένα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις σχετικά με την εξυγίανση και ε, θα συμμετέχουν στις αποφάσεις αυτές και τα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης εξετάζουμε τη δυνατότητα ε, ε, πρόορης εισαγωγής του κοινού προστατευτικού καθεστώτος, δηλαδή νωρίτερα από το 2024. Υπάρχουν ωστόσο τεχνικές προκλήσεις σε αυτό, καθώς το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης προβλέπεται να γίνει αμοιβαίο στα τέλη του 2023. Αυτό σημαίνει πολιτική απόφαση ε, που θα βασίζεται στην ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της μείωση του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα, οι λεπτομέρειες του οποίου ε, προγράμματος τώρα αναλύονται. Τώρα θα στραφώ στο μεταρρύθμιση του μηχανισμού σταθερότητας. Στον Ιούνιο το Συμβούλιο ανέθεσε στο Eurogroup να ε, συντάξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περαιτέρω ε, ανάπτυξη του μηχανισμού σταθερότητας. Ε, αυτό σημαίνει αναθεώρηση ε, προληπτικά μέσα, προστατευτικά μέσα και ρόλο του μηχανισμού σε περιπτώσεις κρίσης καθώς και πρόληψη όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Πρέπει να αποφευχθεί το στίγμα της αγοράς για τις χώρες που ζητούν τη βοήθεια. Είναι σημαντικό να δούμε πώς αυτά τα κριτήρια θα λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό πλαίσιο μάλλον εποπτείας. Ε, ε, η βιωσιμότητα είναι απαραίτητο. Ο ESM θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί το θέμα των, του χρέους στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε λοιπόν τις δυνατότητες διαχείρισης κρίσης αλλά και την πρόληψη ε, αυτής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειάζεται και οικονομική βοήθεια, ας πούμε όσον αφορά την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους. Παράλληλα με αυτή τη συζήτηση, ο πρόεδρος Διακόπτη ζητά από τον κύριο Σεντένο να μιλήσει λίγο πιο αργά για να μπορούν να τον παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ευχαριστούμε. Παράλληλα λοιπόν με αυτή τη συζήτηση γίνεται ε, και η συζήτηση για τη δυνατότητα συλλογικής αναθεώρησης των ρητρών ε, αναδιάρθρωσης, ώστε να μπορεί αυτό να ε, γίνει πιο επικοδομητικά. Θέλουμε επικοδομητικές συζητήσεις και για μια βέλτιστη ε, κατανομή εργασίας ανάλογα με τους θεσμούς και ανάλογα με το τι ανατίθεται σε αυτούς από τις συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο για μας. Να πω και δύο λόγια για το θεσμική μορφή του ESM. Για την ώρα θα διατηρηθεί η διακυβερνητική μορφή. Η ένταξη του ESM σε ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σημαντικός αλλά πιο μακροπρόθεσμος στόχος. Και στρέφουμε τώρα σε έναν άλλο τομέα που ρητά αναφέρθηκε στην δήλωση του Συμβουλίου Κορυφής του Ιουνίου και πρόκειται για το ε, για το ε, Μια πλήρης ε, τραπεζική ένωση θα πρέπει τελικά να ε, προβλέπει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλισης ε, των καταθέσεων. Αυτό το θέμα Ωστόσο, είναι πολιτικό ευαίσθητο γιατί διαφέρουν οι απόψεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις μείωσης κινδύνου που θα πρέπει να τηρούνται. Πολλοί πιστεύουν ότι η πρόοδος θα πρέπει να εξεταστεί επαρκώς τώρα που τα ισοζύγια των τραπεζών βελτιώνονται και που το, οι δέσμοι για τον τραπεζικό τομέα ε, συζητιέται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των τριμερών. Επιτρέψτε μου να στονίσω τη σημασία επίτευξης ε, ε, συμφωνία σε αυτό το τομέα που είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω κατανομή κινδύνων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει τονιστεί από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη στο Eurogroup. Άλλοι θεωρούν πως θα πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση παράλληλα με άλλες συζητήσεις όπως ας πούμε για τη ρυθμιστική ε, εξέταση το, της ε, κρατικής έκθεσης ε, στις τράπεζες και στα ισοζύγια αυτών. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Γιατί είναι σημαντικό για τις αγορές και για τα κράτη. Να πω δύο πράγματα ακόμα για τις ε, ε, δημοσιονομικές δυνατότητες των Ευρωζώνη. Ε, παράδειγμα άλλων ε, νομισματικών ενώσεων όπως η ΕΠΑ και ο πολιτικός ρεαλισμός καθώς και η κατανομή κινδύνου στην ΟΝΕ θα πρέπει να προελθεί από ιδιωτικούς διάβλους και αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση με διασυνοριακές πανευρωπαϊκές τράπεζες καθώς και ε, κεφαλαιακή ένωση. μάλλον ένωση των κεφαλαίων αγορών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και ένα δημόσιο μέσο κατανομής κινδύνου που θα ενισχύει και θα στηρίζει και τον την ιδιωτικό καταμερισμό κινδύνου. Αυτό θα σήμαινε ότι ότι οι χώρες ε, θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν ε, τα δημοσιονομικά τους παρότι αυτή τη στιγμή διαφέρουν πολλοί απόψεις όμως με τον καιρό θα μπορέσουν να βρεθούν δημιουργικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι ανησυχίες υπάρχουν ήδη διάφορες ε, επιλογές αλλά τον Ιούνιο δεν αναφερθήκαμε ακριβώς σε αυτό όμως οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι μεταξύ των θεμάτων που μας ζητήθηκε να συζητήσουμε και το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Επιπλέον το θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το PDP. Ε, να ολοκληρώσω λέγοντας πως είμαι βέβαιος πως το Eurogroup θα μπορέσει να προσφέρει απτή πρόοδο στη διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου. Δεν θα είναι το τέλος ε, των μεταρρυθμίσεων, αλλά θα είναι ένα κρίσιμο ε, στάδιο. Σε ορισμένου τομεί θα χρειαστεί να δουλέψουμε περισσότερο. Προσβλέπω στι δικέ σα κατευθύνσει, ε, τι κατευθύνσει που θα δώσει το Συμβούλιο του ε, Δεκεμβρίου και είμαι στη, βεβαίως διαθέσιμος να κάνω ό,τι μου αναλογεί για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα για να έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική ευρωζώνη που δείχνει πως ξανά και ξανά οι πολίτες ε, ε, έχουν, ε, θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το project. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Σεντένο για την πλούσια και περιεκτική εισαγωγή που μας κάνατε. Πρέπει να πω αναφερόμενος παρατηρήσεις σας για την Ιταλία ότι το παρελθόν σα ω Υπουργού Οικονομικών δείχνει σαφώς ότι είναι δυνατόν σε συνδιαλλαγή με την ε, Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθηθούν ισορροπημένες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές πολιτικές που στηρίζονται και στην δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει ένας και μόνο δρόμος ή ένας οικονομικός κανόνας που υπαγορεύεται αλλά η ευελιξία δίνει τη δυνατότητα των συνδυασμών ώστε να έχουμε κοινωνικές, ε, ε, οικονομικές πολιτικές με κοινωνική διάσταση, με περιβαλλοντική διάσταση. Δεν είναι πιστικό ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να λυθεί το πρόβλημα. Ε, ευχαριστούμε και για αυτά που μας είπατε για τη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ. Εμεί δουλεύουμε πάνω στη δημοσιονομική ικανότητα, έχουμε εισηγητή και ελπίζουμε ότι και το δικό σας το έργο θα συνεχιστεί γιατί είναι ουσιαστικό. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ιδιωτικό επιμερισμό κινδύνου. Είναι δύσκολο αν δεν προχωρήσουμε το αντί την πλήρη οικονομική ολοκλήρωση. Αυτοί που λένε όχι, ότι δεν είναι ώρα για το έντις ακόμα, δεν μπορούν να εξηγήσουν ε, αυτό το όχι. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει και εκείνο να δώσει την συνεισφορά του σε αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο. Ο, πρώτο ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο Ντάριος Ροζάτη για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε μαζί μας ε, σήμερα το πρωί. Πρώτη ερώτηση, το δίλημα μεταξύ επιμερισμού κινδύνου και μείωση κινδυνου κινδύνου. Κάποια κράτη-μέλη είναι υπερχρεωμένα ακόμα, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό και σε περιόδους ε, καλές θετικής οικονομικής συγκυρίας δεν μπόρεσαν να μειώσουν το δίκτυο χρέους και γι' αυτό κάποια άλλα κράτη-μέλη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου γιατί θεωρούν ότι ο κίνδυνος σε κάποιες χώρες είναι πολύ υψηλός και πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε το δίλημα αυτό. Βλέπετε να υπάρχει λόγος για κάποιο περιορισμένο μηχανισμό επιμερισμού του ρίσκου, του κινδύνου αλλά πόσο πιθανό θεωρείται να θεσπιστεί ένα τέτοιο μηχανισμός σε μια κατάσταση όπου όπως είπα έχουμε, πολλές, έχουμε κάποιες υπερχρεωμένες χώρες και μπορεί να υπάρξει και επιβράδυνση το 2019 και σίγουρα το 2020. Για την Ιταλία. Η Ιταλία είναι σε τροχιά σύγκρουσης με την Κομισιόν ε, λόγω του προσχεδίου προϋπολογισμού τους. Είπατε ότι αύριο η Κομισιόν θα εκδώσει γνώμη, αλλά θέλω τη γνώμη τη δική σας και τη γνώμη του Eurogroup σχετικά με το τι μπορεί να γίνει, ώστε να πιστεί ή να ενθαρρυνθεί η Ιταλική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε μέτρα και αποφάσεις που θα μειώσουν την μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη της χώρας και θα επιδεινώσουν τις προοπτικές της. Έχω υπόψη μου την ε, αλλαγή στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Ε, τι μπορεί να γίνει για να πιστεί η Ιταλία ότι πρέπει να σέβεται τους κανόνες και το να διανέμει χρήματα και, και να κάνει λιγότερο ευέλικτη την αγορά από ό,τι είναι τώρα, αυτά δεν είναι σωστά μέτρα για να προχωρήσει η χώρα αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ροζάτη. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να κατανοήσουμε ότι πρέπει να μειώσουμε το κίνδυνο στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη Έχει ήδη μια 20ετή ζωή και εμπειρία μετά τη δημιουργία του ευρώ. Έχουμε και εμπειρία πριν από την επίσημη ε, θέσπιση του ευρώ, αλλά βέβαια είναι σύντομη η εμπειρία αυτή, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Και υπήρξε μία περίοδος κατά την οποία ζήσαμε μία πολύ μεγάλη ύφεση. Και έτσι δημιουργήθηκαν όλες οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί που αναφέρατε. Και η γνώμη του Eurogroup είναι ότι πρέπει να ε, συνδυάσω με τον επιμερισμό και τη μείωση του κινδύνου. Να τα συνδυάσουμε. Ε, και θα πρέπει οι οικονομίες μας να προχωρήσουν σε μέτρα που πολλές φορές μπορεί να είναι και δαπανηρά σε σχέση με το οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτή η απομόχλευση που θέλουμε πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις και σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο και από πολιτικές ε, που θα συνοδεύουν τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια ώστε όλα να εντάσσονται σε ένα, μια συνεκτική δέσμη πολιτικών. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όταν δείτε τους κινδύνους από το Brexit και την οικονομική πολιτική του Τραμπ. Όπως είδαμε πρόσφατα. Πρέπει να φροντίσουμε οι πολιτικές μας να είναι συνεκτικές και συνεπείς στην Ευρωζώνη και η μείωση του κινδύνου σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της. Τώρα για την Ιταλία. Η Ιταλία εντάσσεται σε αυτή την προοπτική. Πρέπει να δώσουμε χρόνο για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε την τελευταία δεκαετία η Ιταλία ε, για να μπορέσουν να οριμάσουν, να δώσουν αποτελέσματα, να ωφελήσουν τους πολίτες. Το Eurogroup στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τη γνώμη της, ε, για το TPP. Και πάλι χρειαζόμαστε έγκαιρα μεταρρυθμίσεις, ε, δίνοντάς τους χρόνο για να οριμάσουν και να αποδώσουν. Αυτό θα ήταν η καλύτερη συμβουλή που θα είχα σε αυτή τη συγκυρία να δώσω στους Ιταλούς. Ευχαριστώ. Υπερβάν Σπερές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε που είστε εδώ μαζί μας ε, στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων. Ε, θα ήθελα ε, να ακολουθήσω την τροχιά της ερώτησης του Δαρίου Ροζάτη ε, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα στο τραπέζι του Eurogroup τα οποία έχουμε εντάξει και εμείς στο πρόγραμμα εργασίας. Θέλω να πω ότι ε, κυρίως η ερμηνεία που ορισμένοι έδωσαν ε, στο Eurogroup ανάμεσα στη μείωση του κινδύνου και τον διαμοιρασμό του κινδύνου. Ναι, νομίζω ότι εάν ρωτήσουμε ε, πώς ερμηνεύει κανείς ε, την, ε, το μοίρασμα του κινδύνου θα έχουμε μεγάλο φάσμα απαντήσεων που θα πηγαίνει από τις τράπεζες μέχρι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί επιμένουμε στη μείωση κινδύνου. Βλέπω τα πρακτικά και την ανακοίνωση τύπου ε, του Eurogroup μετά το πέρας των εργαζιών ε, και λέτε ότι το Eurogroup προτείνει ένα μηχανισμό σταθερότητας και σύγκλησης. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι και πολύ ισορροπημένα. Πρώτα απ' όλα τι θα βάλετε ε, σε αυτό το διαμήρασμα κινδύνου γιατί το backstop το 2024 δεν αφορά ε, ε, ισορροπία λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς εναλλασσόμενες καταστάσεις. Γι' αυτό θέλουμε μια πιο σταθερή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Απαντά ο κύριος Σεντένο. Ευχαριστώ κύριε Μπερέσε. Θα σας απαντήσω στα αγγλικά εάν δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Είναι πιο άνετο για μένα να μην αλλάζω γλώσσες και συνέχεια. Δίκιο έχετε. στη συζήτηση μεταξύ μείωσης κινδύνου και επιμερισμού του κινδύνου και τα σχετικά μέτρα πρέπει να πιέσουμε και προς τις δύο κατευθύνσεις και καμιά φορά δεν φαίνεται να προχωρούμε τόσο γρήγορα ε, στο ένα σκέλος από ό,τι στο άλλο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την καρδιά της Ευρωζώνης. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το φροντίζουμε. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Σε άλλες οικονομικές και νομισματικές ενώσεις αυτό είναι μια πολύ μακρά διαδικασία στην ε, αρχική μου δήλωση ως πρόεδρος του Eurogroup ε, ετώνησα την ανάγκη να προχωρήσουμε με τη σειρά της μεταρρυθμίσεις και να μην περιορίσουμε τη συζήτηση γιατί πολλές φορές ε, εμείς περιορίζουμε τη συζήτηση. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να επιμένουμε, να συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία δημιουργεί εσωτερική εμπιστοσύνη στις οικονομίες μας. Η Ευρωζώνη ε, συνεχίζει τώρα. Έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια δώσει 9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, πράγμα μοναδικό για τις, μοναδική, για τις οικονομίες μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δείχνει ότι ε, πολλά επιτεύχθησαν παράλληλα και με αύξηση μισθών. Είχαμε καλά αποτελέσματα στην Ευρωζώνη. Βέβαια πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι, αλλά και να συνεχίσουμε να πιέσουμε περισσότερο προς τον επιμερισμό του κινδύνου. Η μόχλευση στην οικονομία είναι δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία και θα πρέπει να υποστηριχτεί όμως από τα μέτρα μας. Πρόκειται για μια συνολική προσέγγιση ε, και επαναλαμβάνω ότι ε, οι φιλοδοξίες μας δεν πρέπει να περιορίζονται σε λίγους ε, μήνες. Είναι πολύ σημαντικό και εν ώψη των εκλογών να συνεχίσουμε με μακρόπνο και φιλόδοξο σχέδιο. Ευχαριστώ. Μπέρντ Λούκε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά, κυρία Σεντένο. Για την Ιταλία θέλω να ρωτήσω κι εγώ. Είπατε για την Ιταλία. Είπατε λοιπόν ότι αν η Ιταλία τηρήσει τους κανόνες αυτό θα αποτελέσει βάση για βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή τι ακριβώς έχετε κατά νου, τι να κάνει δηλαδή η Ιταλία ε, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες. Πώς θα δώσει έναυσμα για ανάπτυξη. Τα πολιτικά δεδομένα ε, στην Ιταλία δυσκολεύουν τις μεταρρυθμίσεις. Ε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν κάποια δυνατότητα, αλλά πολλά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αν τηρήσει η Ιταλία τα δημοσιο... τις δημοσιονομικές επιταγές της Ένωσης, ε, πώς θα δημιουργηθεί ανάπτυξη. Λάβετε υπόψη ότι τα τελευταία 15 χρόνια η Ιταλία δεν είχε βιώσιμη ανάπτυξη. Καμιά φορά τηρούσε τους κανόνες, καμιά φορά όχι, τα δοκίμασαν όλα, αλλά αποτέλεσμα δεν βγήκε στην Ιταλία. Οπότε, δηλαδή, τι θα κάνατε εσείς, τι συνταγή έχετε για την Ιταλία, ούτω ώστε βάσιμα να ισχυριστείτε ότι αν η Ιταλία τηρήσει τους κανόνες θα έχει ανάπτυξη. Δεύτερον, αν η Ιταλία δεν τηρήσει τους κανόνες, αν η Ιταλική κυβέρνηση σε αυτή την τροχιά σύγκρουσης με την Κομισιόν και ενάντια στους κανόνες, αν επιμείνει σε αυτή τη θέση η Ιταλία. Αποκλείεται αυτή η Ιταλική κυβέρνηση ή μια μετέπειτα Ιταλική κυβέρνηση να πάρει ε, βοήθεια από τον ESM ε αν υποβάλει το σχετικό αίτημα. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι μια χώρα η οποία δεν συμμορφούται προς τους κανόνες δεν έχει σίγουρα πρόσβαση στην βοήθεια από τον ESM. Μπορείτε να μας δώσετε μια τέτοια υπόσχεση. Ευχαριστώ. Ε, να πω κάτι. Αν δείτε τα δεδομένα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια η Ιταλία είχε ανάπτυξη. Τώρα βιώσιμη, μη βιώσιμη δεν ξέρω. Όχι. Όχι, εγώ δεν έκανα ερώτηση σε εσά. Εγώ ρώτησα τον κύριο Σεντένο και δεν είχε βιώσιμη ανάπτυξη, ξαναλέω, η Ιταλία τα τελευταία 15 χρόνια. Γνώμη σα βέβαια, αλλά πάτε στην Eurostat και θα δείτε άλλα στοιχεία. Ο κύριος Σεντένο για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε ε, Λούκε. Η διαδικασία της πρόοδου είναι μακρόπνοη και μακροχρόνια. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε ε, σαν ε, αγώνα ε, μικρών αποστάσεων. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στη συντάξη, στην αγορά εργασίας, στην Ιταλία. Δεν πάω εγώ να υποστηρίξω σόνι και καλά αυτέ τι μεταρρυθμίσεις ε, αλλά, που, που εφαρμόστηκαν, αλλά αυτέ θέλουν χρόνο. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη χώρα μας κράτησε πολύ. Αρχίσαμε να μεταρρυθμίζουμε το, το 2006 το σύστημα κρατικής ε, ε, ασφάλισης και ακόμα συνεχίζουμε, θέλει χρόνο. Και βέβαια ε, όλα αυτά ε, ε, ωφελούνται λόγω της ένταξης στην Ευρωζώνη, η οποία δίνει σταθερότητα στα νομίσματα, αυξάνει τις αποταμιεύσεις στις χώρες μας, γιατί χωρίς σταθερότητα δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Και πρέπει, πιστεύω, να δούμε και τις προκλήσεις που είναι τα κοινωνικά ζητήματα και που τα ανέφερα στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Οι κυβερνήσεις μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις, να έχουν απάντηση. Ε, δεν πρέπει να είμαστε ανυπόμονοι. Αν γινόμαστε ε, περισσότερο ανυπόμονοι, δεν εξυπηρετεί το γενικότερο σκοπό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πρέπει να συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, να τηρούμε τους κανόνες, γιατί έχουν βιώσιμα δημοσιονομικά και ε, εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι εγώ βέβαια εδώ ως οικονομικό, Υπουργός Οικονομικών της ε, Πορτογαλίας, ε, ορισμένα παραδείγματα έδωσα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ανατρέψουμε το κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης με μια ατζέντα η οποία προωθεί την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και εξετάζοντας θέματα ε, δημοσίων οικονομικών, δημοσιονομικά μέτρα. Όλα αυτά είναι σημαντικά για οποιαδήποτε χώρα και για την Ιταλία για να ξαναγυρίσει σε τροχιά ανάπτυξης όπως, όπως είχαμε πρόσφατα παρατηρήσει στην Ιταλία. Και η ερώτηση η δεύτερη αν μπορεί να βοηθηθεί η Ιταλική κυβέρνηση ενώ θα έχει παραβιάσει τους κανόνες να πάρει βοήθεια από τον ESM Κοιτάξτε πολύ σύντομα να σας πω ότι υπάρχουν κανόνες για αυτό το πράγμα και φροντίζουμε οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για όλους. Υποθέτω ότι ο ESM θα εξακολουθήσει να παίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο που απέδειξε ότι είναι τόσο αποτελεσματικό στο παρελθόν. Όταν έρθει εκείνη η ώρα νομίζω ότι θα παίξει ο ESM βάσει κανόνων. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε κύριε Λούκα ότι ούτως ή άλλως το, το κράτος μέλος ζητά και δεν την ε, προσφυγή και δεν του επιβάλλεται ε, με κανένα τρόπο. Ούτως ή άλλως ε, αν δει κανεί τι αγορέ, ναι, γίνεται μια προσπάθεια από ό,τι φαίνεται <clears throat> για να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να επιβληθεί τίποτα σε μια χώρα, πρέπει να το ζητήσει η ίδια. Ο κύριος Ραμόν Τρεμός παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μάριο Σεντένο, καλώς ορίσατε κύριε Σεντένο στην Επιτροπή μας. Έχω ορισμένε σύντομε ερωτήσεις. Συζητούμε σήμερα ε, το, ε, το backstop για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια Ωστόσο, κάποιοι συντονιστές εδώ δεν καταλαβαίνουν ε, γιατί η οδηγία για τις δευτερογενείς αγορές δεν είναι ακόμα έτοιμες. Ε, πιστεύετε ότι και ο κανονισμός και ε, εμείς πιστεύουμε ότι ο κανονισμός και η οδηγία θα πρέπει να συζητηθούν μαζί. Σας ερωτώ εσάς. Δεύτερον, ενιαίο χρονοδιάγραμμα για όλα τα χρηματοπιστωτικά, για όλες τις πιστωτικές ευρωπαϊκές οντότητες για αυτό το backstop. Ωστόσο, ορισμένα ε, όργανα ε, δεν ε, έχουν την δυνατότητα αυτή. Ερώτηση λοιπόν, δεν φοβάστε μήπως δημιουργήσετε ένα συστημικό σοκ σε κάποιες χώρες γιατί ορισμένες τράπεζες δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το backstop. Για την Ιταλία μια πρόταση. Η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα η οποία είχε πρωτογενέ πλεόνασμα τα τελευταία 20 χρόνια αλλά βέβαια λόγω του υπερβολικού δημοσίου ε, χρέους ε, έχει σημαντικό δημόσιο έλλειμμα κάθε χρόνο. Ο Ευρωπαϊκός ε, Μηχανισμός Σταθερότητας ποιες δυνατότητες θα έχει να χρηματοδοτήσει ενδεχομένως την μείωση των επιτοκίων στην Ιταλία. Απάντηση. Όσον αφορά την οδηγία, για τις ε, δευτερογενείς αγορές ε, όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το επεξεργαζόμαστε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ε, όσον αφορά τις δευτερογενείς αγορές, το τμήμα αυτό δηλαδή του κειμένου υπάρχει μεγάλη συζήτηση από τα κράτη-μέλη. Ε, και ε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον θα υπάρχει υποβοήθηση ε, από τα ACE, αλλά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ουσία είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν μεγάλη μείωση στην Ευρωζώνη. Πρέπει βέβαια να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή της απομείωσης. Και βέβαια και οι δείκτες μείωσης της επικινδυνότητας μείωση του κινδύνου δείχνουν ότι η τάση είναι καλή και σε επίπεδο SSM ε, και στον τραπεζικό τομέα ε, από μόνο του έχουν γίνει πολλές ε, προσπάθειες. Πρέπει να ενδυναμωθεί η διαδικασία με επιπλέον μέτρα. Και οδηγούμε έτσι στην τελευταία σας ερώτηση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, για να τροφοδοτηθεί ε, μια δανειακή κατάσταση πιο ε, βιώσιμη, οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη βεβαίως το πρωτογενές πλεόνασμα αλλά ξέρετε ότι η σχέση ε, εμπιστοσύνης και απόδοσης ε, στην αγορά είναι πάρα πολύ ε, σημαντική και επομένως πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και πώς αντιδρούν οι αγορές και να είμαστε βέβαιοι ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες τελικά γίνονται πραγματικότητα και εκλαμβάνονται με το πραγματικό τους μέγεθος και στις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχουν στρατηγικές ε, βέβαια οι οποίες ξεφεύγουν από τους κανόνες ε, ε, που έχουμε συμφωνήσει όλοι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικέ, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε οι εναλλακτικέ να εντάσσονται στους κανόνες που έχουμε θεσπίσει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίπεδο ε, μικρότερης κατανομής fiscal stance σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι σημαντικό για τις ε, αγορές και είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να στείλουμε στις αγορές και είναι θετικό. Ευχαριστώ πολύ να σου εγώ θα σας ρωτήσω κάτι στα ισπανικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, χθες ε, προχωρήσατε τη συζήτηση για μια εφορολογική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Ε, αυτό μπορεί να είναι ικανοποιητικό, θετικό, αλλά ε, έχουμε μερική την αίσθηση ότι ε, εδώ έχουμε και μία περίεργη άσκηση όπου ναι, ναι, όλοι έχουμε τον προϋπολογισμό, αλλά όταν μπούμε και ωραία και καλά, αλλά όταν μπούμε σε λεπτομέρειες τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία ε, ε, αν πρέπει να υπάρχουν ε, τέτοιε προϋποθέσεις για την δημιουργία μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης, τότε έχουμε ένα είδος ταμείου συνοχής, ας πούμε, και δεν είναι πραγματικός προπολογισμό το ζήτημα και δεν είναι πραγματική σταθεροποίηση. Εσείς ποιον ρόλο θεωρείτε ότι μπορεί να έχει το Eurogroup και επίση όσον αφορά τη διακυβέρνηση αυτή είναι η δεύτερη ας πούμε ερώτησή μου. Ε, εδώ μιλάμε για διακυβερνητική διάσταση και επομένως το εργαλείο αυτό ποιος θα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Θα είναι ε, μικρός ρόλος, θα είναι απομειωμένος ρόλος του, του Κοινοβουλίου ε, και ε, θα είναι παρόμοιος με τον ρόλο του Μηχανισμού Σταθερότητας του ESM ε, ε, το θέμα είναι, ε, θα έχει λοιπόν αυτός ο προπολογισμό θα έχει ή δεν θα έχει σταθεροποιητική ικανότητα και δεύτερον ποιος θα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε αυτό το νέο μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι στα αγγλικά θα σας απαντήσω κύριε Ουρτασούν να υπάρχει συνέπεια σε όλη τη συζήτηση. Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Τονίζω τα εξής πάντως. Χθες δεν βγήκε αποτέλεσμα, τελική απόφαση δηλαδή, σε κανένα θέμα που συζητήσαμε ε, και χθε και στις προηγούμενες συναντήσεις ε, αναφέρομαι, πάει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση το Δεκέμβριο. Αλλά τα θέματα, τα δημοσιονομικά, είναι μακροπρόθεσμα θέματα όπως τα λέμε θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε. Επίσης έγινε χτες μια συζήτηση για το κείμενο Γαλλίας-Γερμανίας. Δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες μόνο, οπότε σίγουρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να το εξετάσουμε. Και αναφερόμενος στη θέση σας θα ήθελα να πω ότι οι φιλοδοξίες γύρω από το τραπέζι διαφέρουν σχετικά με το θέμα αυτό και πρέπει να συγκλίνουμε σε μία θέση κοινή. Ακόμα δεν έχουμε τέτοια κοινή θέση. Οπότε αυτή είναι μία συνεχιζόμενη συζήτηση για μας. Επίσης, πρέπει να εργαστούμε ε, για το, το, σχεδιασμό, το ρόλο του ESM, το μελλοντικό ρόλο του ESM. Το έγγραφο Κομισιόν ESM είναι πολύ ρηξικέλευθο. Όπως είπα και στην αρχική μου δήλωση είναι ένα έγγραφο το οποίο συνάδει απόλυτα με τις συνθήκες. Ε, δεν υπάρχουν κίνδυνοι δηλαδή ε, έλλειψης λογοδοσίας δεν ε, γίνονται τέτοιες προτάσεις από το, την Κομισιόν και τον ESM οπότε από αυτή την άποψη ε, σίγουρα κινούμεθα στο πλαίσιο των εφισταμένων κανόνων και δεν συζητάμε προτάσεις ή θέματα εκτός πεδίου λογοδοσίας των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Πάντα το φροντίζουμε αυτό και πάντοτε το εξασφαλίζουμε. Και για να κλείσω, η δημοσιονομική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Στην ε, ΟΝΕ πρέπει να συμπληρώσουμε τους δημοσιονομικούς μας κανόνες και με άλλα μέσα και μηχανισμούς και αυτό θα κάνουμε στο μέλλον και γιατί σίγουρα οι ανησυχίες που εκφράσατε θα συνεχίσουν να υφίστανται και κατά τη διάρκεια των μελλοντικών συζητήσεων. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στη Μαρίζα Ματίας για την ΚΟΕ, ο Λούντεκ Νίτερμαϊερ, ο αντιπρόεδρος θέλει να ε, ε, θα αναλάβει γιατί έχω κάποια δέσμευση σε σχέση με το Brexit. Σας καλωσορίζω και εγώ. Τώρα η, Μαρία, η Μαρίζα Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Εσείς ε, κύριε Σεντένο διατελέσατε Διατελέσατε υπουργό τη χώρα μα ε, που κατάφερε να αντιστρέψει πολλέ από τι πολιτικέ ε, που επέβαλε η ε, Τρόικα. Αυτές οι πολιτικές αναφίβολα είχαν θετικό αντίκτυπο οικονομικό και κοινωνικό και για τους δημόσιους λογαριασμούς μας. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς Ε, και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ε, στηρίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η οικονομική καταστροφή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Βλέπουμε απειλές ε, στην κυβέρνηση, απειλές και προς την Ιταλική κυβέρνηση, πόσο και αν δεν μας αρέσει, εκλέχθηκε από τους ίδιους τους Ιταλούς δεν θα πρέπει να κάνουμε στους άλλους αυτό που δεν θα θέλαμε να κάνουν σε εμά. Δεν θεωρείται πως υπάρχουν ε, όρια. Δεν μπορούμε όλα να τα δικαιολογούμε ε, στην, στο Eurogroup. Η υπόθεση της Ελλάδας είναι νομίζω η πιο ε, καταφανής. Οι Έλληνες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα υπό την απειλή της ε, ε, ε, αποβολής. Η, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Μιλήσατε για εξαιρετική ανάπτυξη του προϋπολογισμού στην Ελλάδα, αλλά ανάμεσα στο 12 και το 18, 59,6 αυξήθηκε το χρέος, δηλαδή 73% ακόμη και ακόμα 6 πόντους ε, στο 2018 αυξήθηκε το χρέο. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι, τι εννοείται όταν λέτε ότι τήρησε ε, το, τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις. Και υποτίθεται ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα υπήρχε και μια αναδιάρθρωση του χρέους. Θέλω να ξέρω ποια θα είναι αυτή η αναδιάρθρωση του χρέους. Τι σημαίνει ε, ότι δηλαδή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκτός που υποτιμούν τη δημοκρατία υποτιμούν και τα ίδια τους τα λόγια τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά επειδή ε, μιλώ συνέχεια στα αγγλικά. Στην Πορτογαλία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα επιτεύγματα της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια. Και στο Eurogroup και στην Ευρωζώνη θεωρούμε πως πρόκειται για μια διαδικασία όπου πραγματικά ε, ε, έπρεπε να αναφερθεί και να επενεθεί. Ακριβώς ε, γι' αυτό έχουμε τη δημοκρατία, γιατί ακριβώς αποτελείται από εναλλακτικέ και πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τις εναλλακτικέ που υπάρχουν και πρέπει πάντοτε να τις αναζητούμε. Το τι πετύχαμε, το πετύχαμε μέσα στο πλαίσιο των κοινών μας κανόνων. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, ότι ε, το πετύχαμε μέσω της ε, εγχώριας εμπιστοσύνης και της εμπιστοσύνης της αγοράς, ε, που είναι ακόμα πιο σημαντική και δεν θέλω να παραστήσω ότι είμαι εγώ ο, τίποτα το ιδιαίτερο υπουργό Οικονομικών αλλά ε, όντως μπορεί αυτό να ε, θεωρηθεί το παράδειγμα της Πορτογαλίας ως καλό παράδειγμα στην οικοδόμηση της Ευρωζώνης. Το ίδιο για την Ελλάδα. Αυτό που βέβαια μπορούμε να ε, γιορτάσουμε είναι ότι επανήλθε η πολιτική διαδικασία στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική πορεία πριν την κρίση ήταν ε, δημοσιονομικά αβίωτη. Ε, αυτό έπρεπε να γίνει αντιληπτό και να διορθωθεί. Πήρε περισσότερο χρόνο από όσο οποιοδήποτε επιθυμούσε, προσωπικά αυτή είναι η δική μου γνώμη, και συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτή την ε, πορεία Σίγουρα με τα μέτρα υπομείωσης χρέους που, που μελετώνται για το μέλλον και σίγουρα εξετάζοντας τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες της Ελλάδας οι οποίοι βελτιώνονται και ελπίζω πως αυτό θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού εν τέλει. Ευχαριστώ. Και... Δεν μπορούμε να κάνουμε πέντε λεπτές ε, ε, ερωταπαντήσεις γιατί ο χρόνος τελειώνει, γι' αυτό παρακαλώ να είστε πιο, σύντομο, πιο σύντομοι, διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Μπορώ να σας ε, υποσχεθώ ότι εγώ δεν θα ε, σχολιάσω τις υπόλοιπες ε, εκθέσεις. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σεμονόφ. Παρακαλώ σύντομος να είστε. Χωρίς μικρόφωνο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο συνάδελφος Λούκε, θα ήθελα να επανέλθω ε, στην Ιταλία είναι ε, ε, θεμητές οι διεκδικήσεις της Ιταλίας. Στην ε, χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη, όπου ο Μοσκοβισή φαίνεται να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δημοσίων δαπανών. Δηλαδή κάθε ευρώ που δίνεται στην οικονομία, στην αγορά, διευρύνεται και εν τέλει δίνει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στα δημόσια ταμεία οι Ιταλοί τα τελευταία χρόνια σφίγγουν το ζωνάρι όλο και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά ε, τα δημόσια οικονομικά δεν βελτιώνονται λόγω της λιτότητας. Ε, αυτή η ευρωπαϊκή, ε, η ευρωπαϊκή συνταγή με τους κυρίους Ρέντζι και Μόντι δεν λειτουργήσε εδώ. Προβλέπεται πλέον μια ανάκαμψη της οικονομίας με, μέσω της βοήθειας στους φτωχότερου, μέσω της μεγαλύτερης κατανάλωσης των ε, πολιτών ε, και των οικοκυριών και επομένως ε, η αύξηση μπορεί να είναι πολύ καλύτερη. Μετά από την εξυπηρέτηση του χρέους θα μπορούσε να παραμείνει, θα παραμείνει από το 3% το το έλλειμμα στην Ελλάδα ε, ε, είναι γεγονός ότι ε, δεν ελήφθη σωστά υπόψη το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτής της ελιτότητας Στην ετήσια συνάντηση του Παγκοσμίου του, του Νομισματικού Ταμείου στην, στον Παλή αναγνωρίστηκε το λάθος εκτίμησης που έκαναν για την Ελλάδα και αναρωτιόμαστε εάν συνεχιστούν αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι λάθος εκτιμήσεις ε, ε, δεν πιστεύετε ότι τελικά θα υπάρξει έκρηξη εκ των έσω στην, στο Eurogroup. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτά. Απάντηση. Μερικά γενικά σχόλια να σας πω ότι εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σας ε, ότι έχουμε χαοτική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Το αντίθετο μάλιστα, ε, ε, εδώ και 22 τρίμηνα συνεχόμενα έχουμε ανάπτυξη, έχουμε μείωση της ανεργίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα με μικρότερες φορολογικές διασπαθήσεις σε επίπεδο χωρών έχουμε καλύτερο ε, συντονισμό ε, στα πλαίσια ε, περίοδου ανάκαψης. Είναι γεγονός ότι οι δυσκολίες είναι συγκεκριμένες και ότι υπάρχουν δυσκολίες και ότι ορισμένες όντως κάνουν περισσότερο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να λυθούν. Δεν πρέπει να απευθυνόμαστε στο θυμικό και στα συναισθήματα μόνο των πολιτών. Είναι σημαντικό να μιλάμε με λογική και να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο τον οποίο έχουμε ξεκινήσει. Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ε, μέλλον αντάξιο των προσδοκιών μας και των προσδοκιών της κοινωνίας. Και επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τους κοινού μας κανόνες. Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και των αγορών και των πολιτών. Ο Μάρκος Πρέτσα, τελευταίος ομιλητής. Not... Θα μιλήσω γερμανικά. Είμαστε σε φάση ανάκαμψη. Η ανάκαμψη βέβαια δεν ήταν αυτή που ήλπιζαν και ονειρεύονταν πολύ. Πάντως, παρά τη φάση ανάκαμψης, έχουμε και προβλήματα. Τα είπατε κι εσείς εν μέρη. Η Πορτογαλία είναι ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσουν τα πράγματα και πώς μια χώρα μπορεί να ξαναγυρίσει στις ε, κεφαλαίες αγορές που κάποια φάση, σε κάποια φάση ήταν κλειστέ για τη χώρα αυτή. Μιλήσατε και για την Ελλάδα, σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα. Είμαι λίγο επιφυλακτικός εδώ και θέλω να το πω σύντομα γιατί βλέπουμε πάλι συνενώσεις, το παράδειγμα της Τράπεζας Πυραιός και άλλα συγχωνεύσεις. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως στην Ελλάδα βλέπουμε κυρίως ότι η Κομισιόν αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι δέον γενέστε. ε, για τις συντάξεις κλπ. Πιστεύετε ότι οι αγορές θα εμπιστευτούν τελικά στην Κομισιόν ή στον, ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης μιλήσατε και για ε, τους ελέγχους της πολιτικής. Ο έλεγχος της πολιτικής είναι σε χέρια της κυβέρνησης. Αυτό έχει συζητηθεί στο Ευρωζώνη. Δηλαδή, τι προβληματισμός σχετικά με τη δημοκρατία συνδέεται με, αυτή την, αυτό το πέρασμα. Και για την Ιταλία, από το 2000 έχουμε υψηλότερα ελλείμματα από ό,τι βλέπουμε φέτος στην Ιταλία. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι νέα γραμμή πλεύσης της Ευρωζώνης. Δηλαδή η Ευρωζώνη πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον στα θέματα αυτά και είναι απόλυτη προϋπόθεση ούτω ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου να εφαρμοστεί το backstop ε, μετά το 2024. Ευχαριστώ κύριε Πρέτσελ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η Ευρωζώνη είναι μια ομάδα υπουργών οικονομικών και ο ρόλος μας είναι συντονιστικός στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι σημαντικό και για να συνεχίσουμε έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί και ομόφωνα, να παίρνουμε κοινέ θέσεις και αποφάσεις ε, σε σχέση με όλη αυτή τη μακρά διαδικασία ανασυγκρότησης που είναι το ευρώ. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε ανυπόμονοι με τη διαδικασία αυτή. Αλήθεια είναι ότι όταν ε, μας έπληξε η κρίση δεν είμαστε πλήρως έτοιμοι για να την αντιμετωπίσουμε. Από τότε όμως Κάναμε πράγματα. Θεσπίσαμε πολλά μέσα στον τραπεζικό τομέα, στο δημοσιονομικό τομέα, στη, σε, δηλαδή μέσα σε επίπεδο ευρωζώνης, όπως ο ESM, ο Ευρωπαϊκός ε, Μηχανισμός Σταθερότητας. Και Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, αναφέρατε διάφορες ε, περιπτώσεις, πρέπει να συνεχίσουμε να φροντίζουμε ώστε οι πολιτικές που εφαρμόζουμε να είναι βιώσιμες, ε, αξιόπιστες, γιατί η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τις πολιτικές μας και είναι στο χέρι των κυβερνήσεων να αποδείξουν τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία πάντα να το δείχνουν αυτό προφανώς και προς τις αγορές αλλά και προς τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που είσαστε και πολύ ακριβείς στις ερωτήσεις. Αρχίζω με το δεύτερο γύρο. Περιοριστείτε σε ένα λεπτό γιατί αλλιώς δεν θα προλάβει ο κύριος Σεντένου να τα απαντήσει όλα. Ο κύριος Λάγκεν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και εγώ γερμανικά θα σας τα πω. Η αισιόδοξη οικονομική σας πρόγνωση με ενόχλησε λιγάκι. Αναδρομικά, ναι, θετικά 22 τρίμητα, αλλά οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Τα πρώτα ε, ε, προηγούμενα ε, επιχειρηματικά στοιχεία έχουν δοθεί και η θετική σας πρόγνωση έχει προβλήματα και στο Brexit και στην ενεργειακή πολιτική και πολλά άλλα. Για πείτε μου παρακαλώ τα επόμενα τέσσερα τρίμηνα πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Μιλήσατε για, τον ESM. Επίσης, πριν από πέντε χρόνια μας υποσχεθήκατε ότι ο ESM θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Ε, αυτό πάει για αργότερα. Ε, είναι δημοκρατική απάντηση αυτή. Επίσης, η δημοσιονομική ικανότητα. Η δημοσιονομική ικανότητα μπορεί να συζητηθεί, θα συζητηθεί. Τι διαστάσεις πρέπει να έχει για να ε, κάνει όλα αυτά που ελπίζει να κάνει η Ευρωομάδα και δημοσιονομικό πλαίσιο κλπ. Και, και τέλος για την Ιταλία όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έκαναν, ε, εξαιρε... Ε, έκαναν βήματα σύγκλησης με μία εξαίρεση ή την Ιταλία. Και είναι υπερβολικό ότι ο κύριος Μοσκοβισή ε, ε έψεξε εδώ την Ιταλία. Εμείς 10 χρόνια δεχόμαστε η την ιταλια και ειναι υπερβολικο οτι ο κυριος Μοσκοβισσή ε εψεξε εδω την ιταλια εμεις δέκα χρονια δεχομαστε η γαλλια να έχει αυξημένα ποσοστά. Η σκάλα μόμπιλε, ε, ε, ε, μήπως είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει, η οποία παρακολουθεί πληθωρισμό και άλλους οικονομικούς δείκτες. Ευχαριστώ κύριε Λάγγεν. Το Brexit, η Κίνα, το παγκόσμιο εμπόριο, όλα αυτά είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε οικονομικό επίπεδο. Η, η επιβράδυνση που βλέπουμε σήμερα είναι φυσιολογική μετά την ε, αύξηση το 17. Ε, είχαμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο το 17. Οπότε αυτό δεν θεωρούμε εμείς ότι είναι οικονομικό πρόβλημα καθ' αυτό. Εμείς ε, είχαμε βάλει εμπόδια στην οικονομική ανάκαμψη περισσότερα από ό,τι είχαμε φανταστεί. Πάντως η διαδικασία της ανάκαμψης συνεχίζεται και είναι ανθεκτική στα σοκ. Αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι που με κάνει πιο αισιόδοξο αν θέλετε, ε, επειδή αυτό είπατε. Αυτό με κάνει αισιόδοξο για το μέλλον, γιατί μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό μας πλαίσιο με τρόπο τέτοιο, ώστε το τελευταίο να μπορεί να αντέχει τέτοια σοκ. Τώρα για την Ιταλία. Θυμίζω το ύψος του χρέους της Ιταλίας. Είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το έχουμε πρώτο στο μυαλό μας όταν ε, καθορίζουμε πολιτικές δημοσιονομικές για την Ιταλία γιατί το ύψος του χρέους είναι πολύ ψηλό με βάση οποιαδήποτε οικονομικά πρότυπα από όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό δεν μπορούμε παρά να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν πρέπει να φοβάστε για οποιαδήποτε έλλειψη δημοκρατία δημοκρατίας ή δημοκρατικότητα όσον αφορά τις εξελίξεις και το διάλογο και τη συζήτηση. Και μάλιστα και ο ΙΕΣΕΜ μαζί με την ε, Κομισιόν ε, δημοσίευσαν χθες ε, ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται εντός των πλαισίων των ε, συνθήκων. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε ότι θα μπορεί να προκύψει ενδεχομένως οποιαδήποτε εξέλιξη εκτός των κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος ε, Περέιρα από τις, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Μάριο Σεντένο. Θα αρχίσω να, καταρχάς αναγνωρίζοντας ότι το έργο σας ως Πρόεδρο του Eurogroup είναι πολύ δύσκολο. Ε, όλοι γνωρίζουμε πως είναι σημαντικό και επίγουσα μια μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για να προετοιμαστούμε για το επόμενο σοκ. το πολιτικό περιβάλλον δεν θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολο. Ε, έχουμε σύγκρουση δημοσιονομική με την Ιταλία, αστάθεια πολιτική σε κάποιες χώρες και προεκλογική περίοδο και Brexit το Eurogroup θα μπορέσει ήδη το Δεκέμβριο να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και κάποια βήματα για τη μεταρρύθμιση, αν τα καταφέρει αυτό, θα είναι ήδη θετικό το αποτέλεσμα. Κυρίως ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το, προστατευτικό ε, περίφημο καθεστώς ε, για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Ποια είναι η πολιτική σας βούληση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ώστε αυτό το Ταμείο να γίνει πλέον λειτουργικό να τεθεί σε λειτουργία. Δεύτερο, σε, από ποιο σημείο και μετά διατηρείται αυτός ο στόχος της ένταξης του μηχανισμού σταθερότητας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Εάν εδώ μεταξύ υπάρχει χώρος για να ανατεθεί η ευθύνη αυτού, μάλλον για να υποβληθεί αυτή η πρόταση ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα αυτού μέσω μιας συμφωνίας διαθεσμικής στο πλαίσιο μιας διοργανικής συμφωνίας για τα, την ε, λειτουργία και την, το συντονισμό της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Περέιρα. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Έχετε δίκιο ότι βρισκόμαστε σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας το οποίο χαρακτηρίζεται από θετική πολιτικό οικονομικό πλαίσιο και φρέσκους πολιτικούς κύκλους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά σύμφωνα με τα οποία ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στις αρχές αυτού του χρόνου. Όμως τα πράγματα αλλάζουν και προσιάζουμε με προεκλογική περίοδο και ο κίνδυνος που αναφέρατε, ε, ο πολιτικός κίνδυνος ε, όντως ισχύει σε διάφορες χώρες. Υπάρχει όμως μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η σημασία του προστατευτικού καθεστώτος, backstop, Ε, έχει να κάνει με την αξιοπιστία της ίδιας της διαδικασίας εξυγίασης. Ε, δεν μπορεί τέτοια διαδικασία να εφαρμοστεί με συνέπεια χωρίς τη δυνατότητα χρηματοδότησης που μόνο ένα τέτοιο προστατευτικό καθεστώς μπορεί να παρέχει. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη διάσταση της Τραπεζικής Ένωσης. Και ε, ε, είναι επιθυμητή λοιπόν η εφαρμογή αυτού γιατί δείχνει τη δέσμευση των χωρών αλλά θα είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αγορές πως οι ευρωπαϊκές χώρες πραγματικά στηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό αν και πρέπει ακόμα να το συζητήσουμε. να πω δύο λόγια για την ε, λογοδοσία του ESM. Ε, αυτό, επ' αυτό έχουμε εργαστεί στο Eurogroup και νομίζω πως μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Ο κύριος Κίρτσος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το ελληνικό χρέος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αυξηθεί στο 182% του ΑΕΠ στο τέλη του 2018. Αυτή είναι η εκτίμηση του Οκτωβρίου. Ε, η πρόβλεψη του Ιαρινή ήταν 177, κάτι ψηλά. Πώς μπορούμε να συνδυάζουμε λοιπόν αυτή την απόδοση ενώ αυξάνεται περαιτέρω το χρέος. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε ή να σας στείλω κάποιο σημείωμα. Έχει να κάνει με την διαχείριση του ελληνικού χρέους. Το δανεισμού δηλαδή φέτος για να πληρώσουμε τα χρεωστούμενα του επόμενου. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη έχει να κάνει με την τραπεζική κρίση που σοβεί στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί το χρηματιστήριο είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά τις ε, ελληνικέ τράπεζε Έχουν χάσει πάνω από το 50% ε, της αξίας τους από το... και εφόσον δεν μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα ε, δάνεια. Δεν υπάρχουν αρκετές τράπεζες. Αυτή είναι άλλη μια κρίση λοιπόν. Ε, οι δυσκολίες του τραπεζικού τομέα να μην λέμε κρίση, να λέμε δυσκολίες καλύτερα. Έχετε νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες σε επίπεδο Eurogroup. Η ομάδα εργασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Κίρτσο η δυναμική του δημοσίου χρέους πολλές φορές πράγματι είναι εξαιρετικών διαστάσεων και εκθετικές. Πώς αντιμετωπίζουμε με τέτοια δυσκολία. Σταματάμε τη διαδικασία, την αναστρέφουμε και την βάζουμε σε καθοδική πορεία. Οι οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι το πιο σημαντικό είναι ε, ε, όχι τόσο το ύψος, αλλά η τροχιά, η, πορεία του χρέους είναι σημαντική. Όταν αρχίζει να παίρνει καθοδική, να μπαίνει σε καθοδική φάση η καμπύλη του χρέους, τότε βελτιώνονται τα πράγματα. Αυτό πιστεύουμε στην Ευρωζώνη και πρέπει να το, αυτό πρέπει να το καταφέρουμε και στην Πορτογαλία και την Ιταλία και την Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τώρα, σε οικονομική άποψη, το σημαντικό είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας κάθε χρόνο και υπάρχουν μέτρα που έχουν ε, ενσωματωθεί στο πρόγραμμα και εφαρμόζονται τώρα, ούτως ώστε να φροντίζουν ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα μείνουν σε ένα λογικό επίπεδο συμβατό με την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό καθυστερήσαμε την αποπληρωμή ε, μεγάλο μέρος του χρέους και πήγε στο μέλλον. Τώρα επίσης υπάρχει και ένα μαξιλαράκι ε, ρευστότητα που καλύπτει 22 μήνες των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας που θα ε, διαβεβαιώσει τις αγορές ότι η Ελλάδα έχει αρκετά χρήματα ώστε άμεσα να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες αν συμβεί κάποια αναταραχή στην αγορά ή στρέβλωση μη αναμενόμενη να είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τα χρήματα για να ε, γίνει σωστή διαχείριση. Η μόχλευση και η μείωση των κόκκινων δανείων είναι δύσκολο καθήκον και πάλι σημαντικό είναι οι δείκτες αυτοί να πάρουν καθοδική πορεία. Στο βαθμό που βλέπουμε οι δείκτες να μειώνονται μπορούμε να είμαστε ε, ήσυχοι ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες ο Γιάκοπ Φον Βάιτσεκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω για την Ιταλία. Αλλά δεν θα ρωτήσω τελικά γιατί είδα ότι οι απαντήσεις είναι πολύ πιστικές και πράγματι είναι δύσκολη θέση σας ε, ως Πρόεδρου. Τώρα για την δημοσιονομική ικανότητα και την αντασφάλιση, ευρωπαϊκή αντασφάλιση ανεργίας, σε περίπτωση ανεργίας. Όταν ετοιμάσαμε την έκθεση υπερβάνωση εδώ, στο Κοινοβούλιο, δεν μιλήσαμε για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, που υπόκειται βέβαια είναι κομμάτι του ενωσιακού, ένα από τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου προγράμματος κάλυψης της ανεργίας που συζητείτε είναι ότι θα δημιουργούσε μεγάλη σταθεροποίηση και θα έδινε ε, μια διακριτική ευχαίρεια και λόγω του αυτοματισμού του θα μπορούσε, αν είναι σχεδιαστεί καλά, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και θέματα ηθικού κινδύνου και θέματα πολιτικής οικονομίας. Πώς το βλέπετε αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο στα πλαίσια της δημιουργίας μιας σωστής ε, δημοσιονομικής ικανότητας στην Ευρωζώνη. Επίσης, το SBBS, τα SBs που είναι ε, κάτι που μου απασχολεί τώρα είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, που δημιουργεί διάφορες κατηγορίες κρατικών ομολόγων και ως δεύτερο ε, βήμα μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν ως μέσον για την επίτευξη προόδου ούτως ώστε να επιτευχθεί ε, μια αποδέσμευση του πλέγματος που υπάρχει μεταξύ κράτους και τραπεζών. Ευχαριστώ κύριε Φον Είναι πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις σας που απαιτούν βέβαια πολύ μακροσκελείς απαντήσεις από την πλευρά μου κανονικά, ενώ εγώ πρέπει να είμαι σύντομος τώρα. Χρειάζεται σύγκληση, ανταγωνιστικότητα, ευελιξία. Ε, εμείς δεν ε, έχουμε δει ο ναι στον κόσμο που να μην χαρακτηρίζεται από αυτά. Από την αρχή της κρίσης προχωρήσαμε πολύ αναδιαμορφώνοντας το νόμισμά μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και πρέπει να οικοδομήσουμε επάνω στις πρώτες αυτές επιτυχίες. Αυτό που είναι λίγο παράδοξο θεωρώ είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτά που καταφέραμε υπέρ όταν συζητάμε για άλλες μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη και πολλές φορές ε, έχουμε επιφυλάξεις απέναντι στις επιτυχίες μας και αυτό είναι πολύ κακό σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα όταν συζητούμε αυτά τα θέματα που μετριάζουν τον ηθικό κίνδυνο, που δημιουργούν τα σταθεροποιητές, ε, που αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά. Και το μέγεθος. Καμιά φορά φοβόμαστε το μέγεθος των μέσων ή των μηχανισμών. Δεν χρειάζεται να είναι και πολύ μεγάλοι. Απλώς πρέπει να υπάρχουν γιατί έχουν αντίκτυπο ε, στα περιθώρια προσαρμογών που χρειάζεται η οικονομία μας, οι οικονομίες μας που χρειάζονται. Και θα εκπλαγείτε κοιτάζοντας το παρελθόν πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει, τι πρόοδο έχουμε επιτελέσει πράγματα που πριν από 5-7 χρόνια ε, ήταν αδιανόητα, τώρα υπάρχουν. Οπότε ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε όλα τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Μπορείτε να παραμείνετε δύο λεπτάκια ακόμα. Έχω τον κύριο Λούκε, ο οποίο δεν είναι εδώ όμως. Έχουμε ακόμα δύο catch the Εάν και οι δύο συνάδελφοι μπορούν να κάνουν πολύ ε, ε, σύντομες ερωτήσεις, ε, θα, θα υποβάλω εγώ το ερώτημά μου και μετά θα έχουμε και την απάντηση. Ο κύριος Παπαδημούλης πρώτα από την ΓΚΟΕ. 60 δευτερόλεπτα παρακαλώ πολύ. Σημείωσα με ικανοποίηση κύριε Σεντένο τι θετικέ σα δηλώσει για το τέλος των μνημονίων στην Ελλάδα, για την επιστροφή της οικονομίας στην ανάκαμψη και για τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της ελληνικής ε, οικονομίας. Ελπίζω να τις ακούσουν και ορισμένοι στην Αθήνα που επιδίδονται στο σπορ της καταστροφολογίας. Ε, αύριο κατατίθεται η έκθεση της Κομισιόν. Σας έχω ακούσει πριν λίγες εβδομάδες να λέτε ότι με βάση την υπεραπόδοση και με βάση το ότι η πρόσθετη περικοπή των συντάξεων είναι ένα δημοσιονομικό και ένα όχι διαρθρωτικό μέτρο, εάν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, και έτσι λέει το Euro Working Group, για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019, αυτή η περικοπή των συντάξεων δεν είναι αναγκαία. Το ίδιο συνομολογεί πλέον και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Μοσκοβισή μας υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Sorry, we agreed 60 seconds. Uh, next one, 60 Mr. Uh, from non Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Uh, τελευταίος ο μιλήτης. Μια ερώτηση με άλλη οπτική γωνία. Αν τα πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση και τα οποία είναι θηριώδη δεν πιαστούν τα επόμενα χρόνια, αυτό που υποτίθεται ότι συζητάτε για μη περικοπή συντάξεων τι θα γίνει τελικά, θα επανέλθει η περικοπή. Δεύτερον, με τους νέους συνταξιούχους μετά την ψήφιση του νόμου, κατρούγκαλο το ονομάζουμε στην Ελλάδα, του ασφαλιστικού νόμου, που ήδη έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους. Θα παραμείνουν αυτές μειωμένε οι συντάξεις για τους νέους και μελλοντικούς ε, συνταξιούχους. Και τελευταία ερώτηση. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συζητάτε για νέους τρόπους διαχείρισης και την ίδια ώρα φεύγουν και τα τελευταία μέτρα προστασίας της πρώτη κατοικία. 76.000 πληστηριασμοί σπιτιών θα γίνουν το 2019 στην Ελλάδα. Και μιλάτε για κρατικέ εγγυήσει και ομόλογα. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά τα ομόλογα. Τελικά και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, γιατί θα γίνει κρατικό χρέο. Θα μοιράσετε το χρέο ανάμεσα στου φορολογούμενου. Μια ερώτηση ε, στην τροχιά τη ερώτηση του κυρίου Λάγκε. Ε, τα δεδομένα δείχνουν ότι κάποιες χώρες έχουν αρνητική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει επιβράδυνση ή ε, μήπως ε, η πληθυκότητα των δεδομένων δίνει αυτήν την εικόνα. Και τελευταία ερώτηση, έχουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο βουλευτές που επικεντρώθηκαν στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρω... το, το Eurogroup εργάζεται πάντα επί τη βάση των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογήσεων ε, της τωρινής πρόοδου που είναι θετικές μια τέτοια απόδειξη είναι ότι η Ελλάδα δεν έλαβε γράμμα μετά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού. Το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα είναι σημαντικός στόχος και όλα τα στοιχεία για το μέλλον δείχνουν ότι και το 2019 θα έχει την ίδια επιτυχία η Ελλάδα και όλα τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας σε αυτό το πλαίσιο και με την ε, παγρύπνηση της Κομισιόν. Ε, υπάρχει επαγρύπνηση και θα υποβληθεί η έκθεση για, το, για την πρώτη φορά. Τώρα, για την αρνητική ανάπτυξη. Κάποια παραδείγματα αρνητικής ανάπτυξης που είδαμε στα τελευταία τρίμηνα στη Γερμανία ε, οφείλονται σε προσωρινές επιπτώσεις ε, από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία κυρίως. Πρέπει βέβαια να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις διαδικασίες αυτές, αλλά ας μην φοβόμαστε ε, λόγω αυτής της επιβράδυνσης διότι είχε προηγηθεί το 17 πολύ σημαντική ανάπτυξη. Τα μέτρα και πάλι θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης με τρόπο βιώσιμο και αυτό περιμένουμε να συνεχίσει να συμβαίνει ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές στο μέλλον. Ευχαριστώ. Υποσχεθήκαμε να ελευθερώσουμε τον κύριο Πρόεδρο σε 11.30. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Σας ευχόμεθα καλή επιτυχία και ελπίζω η οικονομία να αποδώσει όπως αναμένεται. Θα ξαναρχίσουμε σε ένα με δύο λεπτά. Maybe Pervenche. Let me, let me remind you, we are now starting with point number 15 of Rapporteur Peter Simon. Do we have someone from SND who will take uh, his... Έχουμε κάποιον εδώ από τους σοσιαλιστές, μάλιστα. Τι να κάνουμε, μην περιμένουμε. Okay, because we have, I guess, only a few minutes for, for, for this. Γιατί έχουμε μόνο λίγα λεπτά για αυτό το σημείο. Προβλέψει. 15. Που έχουν γίνει 11. Σημείο 15. Η εφαρμογή των νομικών προβλέψεων της κοινή δήλωση που εξασφαλίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία για τις αποκεντρωμένου τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η ΑΦΚΟ. Ε, η συγητής μας είναι ο κύριος Ζήμαν. Ε, κυρία Μπερές όμως θα παρουσιάσει την γνώμη του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτη φορά ε, σήμερα παίρνω θέση ε, του εισηγητού και γίνομαι σκιώδης. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Τα έκανα μια χαρά και χτες, αυτό το ρόλο τον έπαιξα και επομένως εγώ θα τα πω όμως αγγλικά γιατί έτσι μου είχε αφήσει ο συνάδελφος τις <clears throat> σημειώσεις του. Ο Πίτερ Σίμων λοιπόν είναι ε, συγητή ε, για αυτήν την ε, έκθεση για το κοινοβουλευτικό έλεγχο από των αποκεντρωμένων οργανισμών όπου η ΑΦΚΟ είναι καθήλυν αρμόδια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τον έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών. Η συγητή στην ΑΦΚΟ είναι ο Γεώργης Κόπφιν από το ΕΛΚ. Της 26 Σεπτεμβρίου ο κ. Πίτερ Σάιμον υπέβαλε το προσχέδιο έκθεσης ε, για την ε, ΕΚΟΝ. Ήταν υποχρεωμένος βέβαια ε, να περιοριστεί στο συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Λοιπόν, πέρασε και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Έχουν υποβληθεί 11 τροπολογίες, 3 ε, από το ECR, 3 ε, τροπολογίες από την ALDE, 5 από τον ε, εισηγητή και την υποφαινομένη και μερικές άλλες δικές μου μόνο. 21 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Γενικώ οι τροπολογίες αφορούν ακριβώς τον έλεγχο που θα πρέπει να ε, ε, ασκείται επί των αποκεντρωμένων οργανισμών ε, και αφορούν επίσης εναρμονισμένη διατύπωση με, την, το κύριο κείμενο. μας ενδιαφέρει η εμπλοκή του Κοινοβουλίου, μας ενδιαφέρει επίσης η θέση των ε, υπηρεσιών. Επίσης επικεντρώνονται οι τροπολογίες, τρεις τροπολογίες για την διαφάνεια ως ε, ε, επιτακτικό στοιχείο. Επίσης το γεγονός ότι οτιδήποτε ελέγχεται από το Κοινοβούλιο είναι ε, σημαντικό να συμμετέχει και ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει δίνει προστιθέμενη αξία στο κείμενο και τέλος η θέση του ε, οργανισμού. Δύο τροπολογίες έχουν υποβληθεί από τον Σαλφο σχετικά με την νομοθετική διαδικασία. ε, ε και που σχετίζεται και με τις έδρες των οργάνων και των οργανισμών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσω της συνήθως νομοθετικής διαδικασίας. Επίσης, ε, ε, οι δικές μου τροπολογίες και αυτές του Πίτερ ε, Σέιμον αφορούν τις προθεσμίες, αφορούν τις κοινές εγκαταστάσεις, αφορούν την αποτελεσματικότητα, τη λογοδοσία ναι, καλύτερη αποδοτικότητα για τον προϋπολογισμό και βεβαίως ακεραιότητα, διαφάνεια και προστασία συμφερόντων των εμπλεκομένων. Θα πρέπει οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου να ε, καλύπτονται πάντοτε και οι έδρες ε, των οργάνων θα πρέπει να ε, δίνουν την δυνατότητα για κοινή διοικητική στήριξη και κοινέ υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Έχω και μία τροπολογία την οποία έχω υποβάλει μόνη μου στην τροπολογία αυτή ζητώ από, το, από την Κομισιόν να κάνει περιστατωμένη ανάλυση για την εφαρμογή της κοινή δήλωσης και της κοινή προσέγγισης 10 Ιουλίου του 2012 κτλ. λοιπά και να προδιορίσει την προσαναθεώρηση και εφαρμογή διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω ό,τι αφορά στοιχεία που σχετίζουν με τη δομή και τη διακυβέρνηση και αν οι διατάξει αυτέ είναι αρκετά ευέλικτε να καλύπτουν τον διαφορετικό χαρακτήρα των οργανισμών. Επίση, όσον αφορά και την επόμενη τροπολογία, ο εισηγητή θεωρεί ότι θα πρέπει ε, να ε, ληφθεί υπόψη πάντα με σεβασμό των αριθμών των χαρακτήρων που επιτρέπονται. Σε αυτή την περίπτωση ευχαριστώ. Δεν έχουμε και πολλούς βουλευτέ εδώ. Δεν έχουμε και κανέναν ε, σκιώδη. Θέλει να μιλήσει κάποιο από το ΕΛΚΑ. Όχι. Θέλει να μιλήσει κάποιο άλλο γενικά. Όχι. Α, ήρθατε κύριε Πίρινγκ. Ίσα ίσα ήρθατε έτσι ώστε να μας δώσετε την άποψη του ECR. Όχι από το ECR, από το Άλντε. Συγγνώμη, κάνω λάθος λέει ο Πρόεδρος. Thank you very much for waiting. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με περιμένατε, λέει κυρία Βίρινγκ. Έχω κάποιες ε, τροπολογίες, οι οποίες ε, κατά την άποψή μας είναι σημαντικές αλλά υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες ε, όσον αφορά την γνωμοδότηση αυτή που αφορούν πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά ε, ε, σημεία. Πρέπει να υπογραμμιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας και του τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με το πώς θέλουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία και την λειτουργία των αποκεντρωμένων οργάνων και οργανισμών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον ότι είναι σημαντικό να ε, ε, δίνουμε την ε, δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλλουν θετικά. Ιδίως όσον αφορά το Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία, κυρίως στη φάση ανάμεσα την γενή και τη δευτερογενή νομοθεσία. Τέλος, ε, ε, το μήνυμά μας προς το Συμβούλιο είναι ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ε, τον ίδιο ρόλο με τους υπολείπους στην απόφαση περιεδρών. Είμαστε το, ο οίκος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και επομένω είναι απολύτως θεμητό το αίτημά μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία ε, Βίντρικ που ήρθατε. Α, θέλει κάποιος να μιλήσει, παρακαλώ, με μικρόφωνο. Το πρόβλημα με αυτές τις αποκεντρωμένες ε, ε, υπηρεσίες και οργανισμούς ε, είναι ότι τίνουν να αποκτήσουν τρομερή εξουσία, λέει ο κύριος Ντάτμοθ. και αυτή η εξουσία δεν υφίσταται ικανό έλεγχο. Εκεί είναι το έλεγχο, γιατί ε, είναι ένα πρόβλημα με τις αποκεντρωμένους οργανισμούς. Δημιουργείται ένας αποκεντρωμένος οργανισμός και σιγά σιγά ε, αποκτά μεγάλη εξουσία. Είναι σημαντικό λοιπόν να ελέγχονται, να υφίστανται διαδικασία λογοδοσίας αυτοί οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και ο, ο προφανής ελεγκτής πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η προλαλήσα σας συνάδελφο, πρόεδρο. Και εγώ ε, συμμερίζομαι την άποψή σας ότι το γεγονός ότι οι οργανισμοί είναι αποκεντρωμένοι ε, δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν θα πρέπει να ελέγχονται. Πολύ ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, θέλετε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια, ναι. Ναι, νομίζω ότι ένας από τους κύριους λόγους, κύριε Μπερέσε, που συζητούμε τη γνωμοδότηση αυτή είναι για αυτή τη ε, μεγάλη συζήτηση που έλαβε χώρα ε, ε, σχετικά με την αλλαγή έδρας της, του Οργανισμού Φαρμάκων. Και έχει πάρα πολύ δίκιο ο κύριος Ντάρτμουθ σε αυτό που είπε, ότι δηλαδή είναι σημαντικό να ασκούμε την ε, εξουσία και αρμοδιότητα συναπόφασης και σε αυτές τι περιπτώσεις, όχι μονάχα σε περίπτωση μετεγκατάσταση, γιατί δεν θα έχουμε και τόσε συχνέ μετεγκαταστάσει, αλλά και όσον αφορά την έδρα των ε, οργανισμών. Και είναι πολύ έγκαιρη αυτή η συζήτηση, γιατί ε, έχουμε και αυτήν, την, αυτόν τον οργανισμό τον οποίο ασχολείται και η Επιτροπή ΕΜΠΛ σχετικά δε με την ε, λογοδοσία των οργανισμών βεβαίως είναι εξαιρετικά ε, κρίσιμο σημείο και πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αλλά το τελευταίο σημείο το οποίο ανέφερα σε σχέση με, τον, με τη δικιά μου τροπολογία, εάν δείτε την ε, δήλωση που έλαβε χώρα το 12 ε, θα διαπιστώσετε ότι έχει πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις ε, για το προφίλ και τη διακυβέρνηση, τον ρόλο των οργανισμών και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί καμιά φορά μπορεί να μην είναι και fit for purpose για να καλύψουν ε, τον τόσο ε, ε, το τόσο πολυσχηδές πεδίο το οποίο εμείς καλύπτουμε κάτω από τους οργανισμούς αυτούς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η ψηφοφορία θα γίνει 21-22 Ιανουαρίου. Αυτό είναι το σχέδιο προς ώρας. Ολοκλώσαμε το σημείο 15 και δεν θα ανοίξω το σημείο 16. Α, ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη είναι εδώ, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα του δώσω μάλιστα και την θέση της ε, ε, Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε με την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μία εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Προχωράμε στο σημείο 16. Μία από τις δύο νομοθετικές προτάσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα. Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Πριν δώσω το λόγο πρώτα στην Έσθερα, θα αναφερθώ σε κάτι που δεν αναφέρεται στην ουσία, στην οποία θα αναφερθώ μετά, αλλά στο θέμα της δέσμης. Εμείς δεν ε, δουλέψαμε τις δύο προτάσεις με τον ίδιο ρυθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη δεύτερη την έχουμε εγκαταλείψει. Θέλουμε να ε, ολοκληρώσουμε και τις δύο εδώ λάβαμε υπόψη την καλή δουλειά του Συμβουλίου ως γενική προσέγγιση, οπότε είδαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Τον προστατευτικό, προληπτικό καθεστώς το επιταχύνουμε και στο δεύτερο πάμε με κανονικό ρυθμό και ο στόχος είναι να ολοκληρώσουμε και τις δύο προτάσεις και έτοιμες για να τεθούν σε ισχύ. Ε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και το Συμβούλιο θα μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά, δεν είναι όλα στο χέρι το δικό μας, αλλά κάποιοι σκιώδεις έθεσαν σχετικά ζητήματα. Το μήνυμα είναι ότι δεν εγκαταλείπουμε το άλλο, επιταχύνουμε αυτό γιατί υπήρχαν οι δυνατότητες να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και θα ήταν λογικό αφού ε, συνεχίζουμε και το άλλο τραπεζικό πακέτο να ε, συντονίσουμε τις δύο προτάσεις στα δύο μέρη. Οπότε αυτό είναι λογικό και έτσι εξηγείται η επιτάχυνση. Και η οδηγία είναι σημαντικό κομμάτι της δέσμης. Οπότε μετά από αυτή τη γενικότερη διευκρίνηση δίνω το λόγο στην Έστερ για να αρχίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και το συνεισηγητή μου. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε κοινή θέση με δυο συνεισηγητές. Αυτό σημαίνει ότι η περισσότερη δουλειά γίνεται εδώ στην Επιτροπή. Ήδη ε, έπρεπε να καταλήξουμε σε μια θέση πριν αρχίσουμε να γράφουμε την έκθεση. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Θα ε, λύσουμε και κάποια θέματα που έχουν μείνει μετά την τελευταία οικονομική κρίση. Υπάρχουν ορισμένες αρχές και στόχοι που είχαμε ιδιαίτερα μετά το Συμβούλιο και τη γνωστή θέση του. Πρώτον, θέλαμε να είμαστε γρήγοροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι φάκελοι θα επιβράδυναν, αλλά εδώ χρειαζόταν επιτάχυνση. Η συμφωνία μας επίσης σημαίνει ότι ελπίζουμε να μπορέσουμε να παραδώσουμε τα αποτελέσματα σύντομα, να δώσουμε ένα μήνυμα πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Ταχύτητες είναι σημαντική, αλλά και ο ρεαλισμός. Είμαστε κοντά στο κείμενο του Συμβουλίου για να βρούμε κοινό έδαφος πιο εύκολα. Είμαστε και φιλόδοξοι. Στο τέλος των μακρών συζητήσεων ε, είχαμε ε, για όλες τις κατηγορίες ε, κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων απαντήσεις οι, όλες οι πολιτικές ομάδες ήθελαν να μην περιπλέξουμε πολύ το σύστημα και όταν έχουμε λίγες κατηγορίες, μόνο τρεις, έχουμε ένα απλό σύστημα και έχουμε μια βασική αρχή ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε πιο ήπια καμπύλης για τα προηγούμενα χρόνια ε, λαμβάνοντας έτσι υπόψη κάποιες ανησυχίες των εμπλεκομένων και των πολιτικών ομάδων, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερο κίνητρο ε, πώλησης ε, ώστε τα ανοίγματα να μην μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε δει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες αυτό εξαρτάται από τις τροπολογίες που θα δώσετε ή δεν θα καταθέσετε ε, για ε, ίσως ε, κάποια αναστάτωση στις δευτερογενείς αγορές, κάποια προβλήματα εκεί. Το άλλο είναι αν θα περάσουν κάποια μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλο πιστοτικό ίδρυμα. Δεν είμαι και πολύ υπέρ, αλλά εξαρτάται και από την αξία του δανείου. Θα περιμένουμε εδώ να δούμε τι θα προκύψει από τη συζήτηση εδώ και μετά τις τροπολογίες. Για το μέλλον το θέμα του στόκ των μη εξυπηρετούμενων παραμένει. Εδώ θα πρέπει να είναι και η οδηγία φιλόδοξη για να λύσει αυτά τα θέματα και ε, έγινε και μια σχετική ερώτηση στον πρόεδρο του Eurogroup. Και εσείς θα πείτε για το χρονοδιάγραμμα κύριε Πρόεδρε ακριβώς τι προβλέπετε, ποια, ποιο είναι το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα τις επόμενες εβδομάδες. Φιλόδοξο είναι όντως, ε, αλλά Πολλέ φορέ η Επιτροπή μας κατηγορήθηκε ότι δεν κινείται αρκετά γρήγορα. Τώρα μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και α το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ που είσαστε πολύ αποτελεσματικοί. Χρησιμοποιήσατε λίγο παραπάνω από το μισό χρόνο που είχατε, αλλά αφού τα είπατε όλα ωραία, γιατί όχι και συμφωνώ εγώ με τη συνεισηγήτρια δεν ήταν εύκολα όλα αυτά γιατί είχαμε αρχικές διαφορές αλλά νομίζω ότι το κείμενο και θα ακούσουμε σχετικά τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες σας αλλά όπως είπε και η Έστερ το κείμενο είναι φιλόδοξο, απλό, ισορροπημένο και πραγματικά ε, προβάλλει και προτείνει ένα μέτρο υποχρεωτικού προληπτικού προστατευτικού καθεστώτος για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που είναι κάτι που διαφέρει από την αντιμετώπιση κατά τράπεζα. Είναι ένα μέτρο στεναρό θα έλεγα και ήταν σημαντικό να θεσπιστεί αφενός για να ε, διευρυνθεί ε, και ο, και κίνδυνος ε, αλλά και να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες πτωχεύσεις δηλαδή μιμιέ κλπ. Βρήκαμε λοιπόν μια λύση που αποφεύγει τους κινδύνους αυτούς με μια εξαίρεση που την ανέφερε ήδη η Έστερ και θα πω και εγώ το θέμα των δευτερογενών αγορών, κάποιων δηλαδή παικτών στην ε, δευτερογενή αγορά. Πάντως ε, γενικά η πρόταση είναι ισορροπημένη και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Αυστριακή Προεδρία και το Συμβούλιο γιατί μπορέσαμε να βασιστούμε σε εξαιρετική δουλειά που έγινε και στο Συμβούλιο που έφτασαν σε συμβιβαστική λύση με ομόφωνη στήριξη και η πρότασή μας, οι προτάσεις μας είναι μια παραλλαγή, αν θέλετε, του κειμένου του Συμβουλίου. Αυτή είναι η βάση και περιλαμβάνουν πολλές διατάξεις από το Συμβούλιο σχετικά κυρίως με την απλούστευση και επίσης όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ως πυλώνα 1. Υπάρχει και ο πυλώνας 2. Η λίγο μακρότερη περίοδος για να φτάσουμε σε πλήρη αξιολόγηση είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει ο πυλώνας 1 και μετά υπάρχει και η δυνατότητα του πυλώνα 2 για να προχωρήσουμε γρηγορότερα και πιο σκληρά και εκεί θα υπάρχει προσέγγιση κατά τράπεζα και κατά δάνειο. Οπότε μπορεί να μην είναι αυτό ακριβώς που θα είχα κάνει εγώ, ε, αλλά αντιμετωπίζεται το πυλώνας 1 και 2 είναι μακρότερη η περίοδος για την αυτόματη ε, ρύθμιση και υπάρχει και η δυνατότητα να ε, χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα το πυλώνας 2 και δίνουμε τρία χρόνια χρόνο για πλήρη κάλυψη και όταν βλέπετε 0-0 μετά από ένα-δύο χρόνια δεν σημαίνει ότι είναι 0. Σημαίνει ότι είναι το... Υπάρχει δηλαδή η λογιστική κάλυψη. Υπάρχει κάλυψη η οποία διέπεται από τους κανόνες λογιστικής. Οτιδήποτε είναι πέρα από τους λογιστικούς κανόνες είναι αυτό που προσφέρει ο, πιστοληπτικός, ο προληπτικός προστατευτικός μηχανισμός ή το καθεστώς. Και έτσι έχω μέρο 100% μετά από τρία χρόνια. Ε, ακολουθήσαμε το Συμβούλιο που κάνει αυτή την ε, διαίρεση ε, σχετικά με την κάλυψη από περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή άλλα. έχουμε και πρόβλεψη για μικρότερη πρόβλεψη, όχι όμως όταν πρόκειται για ε, κίνητα περιουσιακά στοιχεία. Εκεί χρειάζεται λίγο, περισσότερη, ε, λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, το, ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος χρόνος είναι τα σημαντικά χρόνια. Εκεί θα αποφασίσουμε τι θα γίνει με το μη εξυπηρετούμενο. Και αν δώσουμε το λάθος κίνητρο, δεν μπορούμε να σώσουμε την εταιρεία που θα μπορούσε να σωθεί και να κρατήσουμε σε αποδεκτά επίπεδα το χρέος, το δάνειο. Πρέπει να υπάρχει μία κάλυψη η οποία σίγουρα θα παρέχει ένα δίκτυο ασφαλείας, αλλά αν πάτε πιο μακριά, στον τρίτο, τέταρτο ε, να υπάρχει ε, πρόβλημα. Μετά η καμπύλη επιταχύνεται και από τη μία πλευρά ε, αποφεύγουμε το αντίθετο κίνητρο. Τα δύο κίνητρα συνδυάζονται με το σωστό τρόπο και με την καμπύλη που προτείναμε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά για τα άλλα θέματα γιατί νομίζω ότι είναι και προφανή αν θέλετε. Τονίζω ένα μόνο αυτό που δεν είχαμε χρόνο για να βρούμε κοινή λύση και το αφήσαμε κάπως ανοιχτό και που αφορά τους παίκτες που έχουν ρυθμιστεί ενώ είναι τράπεζες, ενώ άλλοι παίκτες στην αγορά που δεν έχουν ρυθμιστεί είναι στην δευτερογενή αγορά. Μπορούμε να βρούμε μια λύση που δεν θα τιμωρεί υπερβολικά αυτούς τους ε, δρόντες στην αγορά σε σχέση με τους μη τραπεζικούς. Γιατί αλλιώς ε, μπορεί να ε, προτιμήσουμε άλλους χρηματοπιστωτικούς παράγοντες που δεν υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανόνες. Είναι σημαντικό να είναι ισότιμοι κανόνες του παιχνιδιού και σημαντικό είναι να μην έχουμε αρνητικά κίνατρα. Ε, όταν είναι βιώσιμη η εταιρεία και μπορεί να χρηματοδοτηθεί είναι σημαντικό να μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Ε, και ε, αυτά, αυτά προβλέπονται και στα, για να αντιμετωπίσουμε και τα Gone Concern Capital. θα λάβουμε υπόψη μας και τις ανησυχίες σας και τις τροπολογίες σας για να βρούμε μια ισορροπημένη λύση σε αυτό το ανοιχτό ζήτημα. Μπέρντ Λούκε για το ECR και τον Σάντερ. Ευχαριστώ. Ανέλαβα την έκθεση από τον Σάντερ Λούνς, ο οποίος έγινε υπουργό. Οπότε δεν θα μιλήσω τόσο για λογαριασμό του, αλλά για δικό μου λογαριασμό, γιατί είμαι ο νέος Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για την προκαταρκτική εργασία. Ήδη ακούστηκαν πολλά και σημαντικά. Εγώ εστιάζω στο τελευταίο θέμα που έθιξε ο Ρομπέρτο, δηλαδή ε, επιπτώσεις στην ε, δομή της αγοράς. Να προσέξουμε αν αγορές που δραστηριοποιούνται στη δευτερογενή αγορά θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες ρυθμίσεις όπως και οι τράπεζες ε, στην πρωτογενή αγορά. Ε, μπορεί να θέλουμε να αποφύγουμε στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζών που θα έβλαπτε τις bad banks και πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι δεν το θέλουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να πάει υπερβολικό κομμάτι από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον μη ρυθμιζόμενο τομέα αλλά πρέπει να προσέξουμε αν ε, υπάρχουν, αν δημιουργήσουμε κανόνες ε, εξαιρέσεις ε, γιατί που δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες στη δευτερογενή αγορά να σταθμίζουν και τα, τα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με χαμηλότερες προϋποθέσεις σχετικά με την επάρκεια κεφαλαίων σε σχέση με την πρωτογενή αγορά, τότε θα υπάρξει στρεβλωτικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει τα πακέτα των NPL να ε, πηγαίνουν και να έρχονται και μετά να καταλήξουν στην αρχική τράπεζα. Είναι ένα σύνθετο καθήκον αυτό, όπου ακόμα δεν, έχει, δεν διαφαίνεται ε, οριστική λύση. Θα ε, το, τα κοιτάξω όλα αυτά, θα καταθέσω και σχετικές τροπολογίες και ελπίζω να βρούμε καλή λύση γιατί θέλουμε μια στεναρή αγορά για τα NPLs που δεν θα ε, μένει ε, ε, αυτό το θέλουμε όλοι. Περιορίζομαι αρχικά σε αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρεμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, οπότε να σας συγχαρώ. Γιατί εγώ Ήμουν προβληματισμένος για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος της θητείας. Η φιλοδοξία των μικρότερων ομάδων είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία, να έρθουμε δηλαδή και να πούμε ότι κάναμε κάτι χρήσιμο. Έχουμε μέχρι την Παρασκευή να υποβάλουμε τροπολογίες, ε, οπότε θα δραστηριοποιηθούμε στην ομάδα μου για να πούμε τη γνώμη μας και θα έρθουμε στη συζήτηση σε επικοδομητικό πνεύμα για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το τελικό αποτέλεσμα για να φτιάξουμε ένα νομοθετικό πακέτο. Να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας ε, τι πιστεύετε για την πιθανότητα επανεξέτασης για τη συμπερίληψη όχι μόνο τραπεζών σε αυτή την νομοθεσία, αλλά και άλλων δημοσιονομικών οργανισμών, μεγάλων οργανισμών. Και τι πιστεύετε για την πιθανότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Τραπεζών να μπορεί να βοηθήσει ε, κατευθυντήριες γραμμές για να τους ε, καθοδηγήσει στο να δημιουργήσουν backstops. Ε, βεβαίως ε, μπορεί μία αποδοτική έκθεση τελικά να καταλήξει να μην είναι αποδοτική θα πρέπει να καλύπτονται μέχρι το 80% όπως λέει η Κομισιόν. Αυτό είναι θετικό για μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο και το ανέφερα και στον Υπουργό Σεντένο. Συμφωνούμε πως οι μεγάλοι οργανισμοί θα πρέπει να οικοδομήσουν ε, προληπτικές, ε, ε, προληπτικά καθεστώτα, αλλά στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικά δημοσιονομικά συστήματα με διαφορετικά χαρτοφυλάκια μη αποδοτικών δανείων. Άλλοι, έχουμε, άλλοι έχουν backstop, άλλοι δεν έχουν. Εφόσον λοιπόν έχουμε νομικά πλαίσια που είναι συμπληρωματικά για τα ε, MPL, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να έχουμε μια γενικευμένη προσέγγιση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι καρποφόρα η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές και τους συναδέλφους. Ε, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία, ένα σχέδιο έκθεσης και συμφωνούμε για πολλά από τα σχόλιά σας. Ωστόσο θα πρέπει να πω ότι ολόκληρη συζήτηση για τη αυτού του χρονικού πλαισίου για τις διατάξεις αυτές είναι απογοήτευση. Μιλάμε για εννέα χρόνια ώστε οι τράπεζες πλήρως να καλύψουν τα μη αποδοτικά δάνεια. Ε, τα μη ε, ασφαλισμένα MPL θα έπρεπε κανονικά να καλύπτονται μετά από τρία χρόνια, αν και δεν ε, στηρίζονται από κανένα collateral. Αυτή δεν είναι αποδεδειγμένη προσέγγιση και δεν οδηγεί σε μείωση κινδύνου που πρέπει να επιτύχουμε στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ειδικά ισοζύγια. Ε, και ε, το Κοινοβούλιο στο σχέδιο έκθεσης προτείνει ακόμα μεγαλύτερη αποδυνάμωση από αυτό που συζητείτε στο Συμβούλιο που ε, συζητιέται επί τη βάση μιας αδύναμης προσέγγισης από πλευράς της Κομισιόν και αυτό είναι ακόμα πιο αληθές όταν συγκρίνουμε τις επιλογές που έχουμε επιτάπητο με τους κανόνες που ήδη εφαρμόζονται στη ΣΥΠΑ το ρυθμιστικό πλαίσιο και το λογιστικό πλαίσιο τον είπα, απαιτεί την ε, αντασφάλιση των ε, collateral έξι μήνες μετά από την ταξινόμησή τους ως μη ε, αποδοτικά. Έξι μήνες μόνο έναντι εννέα ετών που θα έχουν τα, οι τράπεζες οι ευρωπαϊκές για να στηρίξουν τα MPL. Στην έκθεση περί MPL το Σεπτέμβριο του 2018 φαίνεται σαφώς πως το αποτέλεσμα της αυστηρής ρυθμιστικής αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων στην, στην, στη ΣΥΠΑ είναι η θετική. Οι Αμερικανικές τράπεζες πολύ πιο γρήγορα μείωσαν αυτά τα δάνεια ε, ενώ η διάθεση αυτών των δανείων έφτασε σε αιχμή μετά από την ε, ύφεση. Ενώ ο όγκος αυτών το, στα τέλη του 2016 στην Ευρώπη ήταν μεγαλύτερος από αυτόν τον όγκο το 2009. Και ξέρουμε ότι εδώ εξαρτώμαστε περισσότερο από τις τράπεζες από ότι στο αμερικανικό σύστημα. Η σύγκριση ωστόσο είναι πολύ εντυπωσιακή. Η εμπειρία από ό,τι είπα δείχνει πως οι τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν σκληρούς κανόνες. Εμείς ως πράσινοι προτιμούμε να είμαστε λοιπόν ε, πιο αυστηροί όσον αφορά το προληπτικό προστατευτικό καθεστώς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ένα μέγα πρόβλημα ε, το οποίο δεν αναφέρουμε. Εγώ θα πρέπει να το κατονομάσω, να πω ότι χωρίς σημαντική μείωση κινδύνου ποτέ θα φτάσουμε σε ένα πλαίσιο ε, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης ε, Καταθέσεων που θα προσφέρει την ίδια προστασία για όλους τους καταθέτες στην Εύρωση και ούτε το δημοσιονομικό προστατευτικό καθεστώς για το ε, ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Κάτι τέτοιο θα εμποδίζει την Τραπεζική Ένωση και τη συμπλήρωση αυτής από ένα τρίτο πυλώνα. Το να έχουμε ισχυρότερο πλαίσιο για το ευρώ σημαίνει σκληρή γραμμή όσον αφορά το προληπτικό προστατευτικό καθεστώς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και ε, Βεβαίω σημαίνει κάτι τέτοιο ότι χρειάζονται και ελάχιστες προδιαγραφές για ε, τις ε, πιστοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν θα ωφελήσει σε τίποτα ε, να χάνει ο κόσμος τα σπίτια του ή τις μικρές επιχειρήσεις ε, από την Τέσσα, Σαν Πάολο και ε, διάφορα banks και όλες αυτές τις ε, δομές θα πρέπει να προστατευτούν οι καταναλωτές μέσω μιας τέτοιας οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό να μην δεχτούμε αυτό το αδιέξοδο για την οδηγία στο Συμβούλιο, αλλά να προχωρήσουμε με τον κανονισμό και την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους ε, συνεισήγητές γιατί είναι πολύ καλό το προσχέδιο της έκθεσης τους. Ε, το χρονοδιάγραμμα είναι ικανοποιητικό. Ε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την, με την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων. Το, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι να έχουν καλύτερη προστασία όσο γίνεται περισσότεροι κάτοχοι. Επίσης μία ρήτρα ε, στα, ε, ε, στα δάνεια έτσι ώστε να δίνει ο καθένας την σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την μεταπόληση σε φαντ. Ε, ο κανονισμός αυτός ε, είναι ικανοποιητικός. Ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και άλλα αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες αλλά θα πρέπει να αναφέρονται και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία που παρουσιάζεται έτσι ώστε ε, να είναι ε, υποχρεωτική η αναγραφή όλων των ε, υποχρεώσεων σε σχέση με τα στεγαστικά ε, δάνεια και σε σχέση με τη δυνατότητα απόλυσης κλπ. Επίσης ε, θα ήθελα να δω ε, να γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι δεν θα είναι πάντα ανάλογα τα επιτόκια ανάλογα με την χώρα και βεβαίως να δούμε ιδιαίτερως τα στεγαστικά τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης καθώς επίσης φυσικά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να είναι πολύ πιο ξεκαθαρισμένες οι προϋποθέσεις και οι όροι βάσει των οποίων θεωρείται ένα δάνειο εξυπηρετούμενο ή όχι και αυτό ε, ανάλογα και με την γενικότερη νομοθεσία της χώρας. Ε, εμείς νομίζουμε ότι μέσω αυτού του κειμένου μπορούμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με την εποπτεία και τη ρύθμιση. Ευχαριστώ. Ο Μάρκο Βάλι δεν είναι εδώ ούτε κάποιος άλλος συνάδελφος από την ΕΝΕΦΕ ή από την EFDD. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι. Άρα να κάνουμε τα τελικά μας σχόλια. Έστερ, ναι, ευχαριστώ συνάδελφοι. Σύντομος αλλά ανανεωτικός έτσι γύρος οι πράσινοι φαίνεται να έχουν ακόμα πιο ε, αυστηρή προσέγγιση από ότι οι φιλελεύθεροι. Άρα εγώ είμαι πιο κοντά στους πράσινους ε, παρά στους ε, φιλελεύθερους. Το αμερικανικό σύστημα και οι έξι μήνες που ανέφερα στην πρώτη μου συζήτηση, στην πρώτη συζήτηση που είχαμε εδώ, είναι πραγματικά πολύ θετικό στοιχείο μουσική στα αυτιά μου. Έχουμε και τον κύριο Λούκα και όλοι μαζί θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ε, μια πάρα πολύ να δημιουργηθεί θα μπορούσε μια πολύ ικανοποιητική συμμαχία μικρών ομάδων. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να το πούμε σαφώς. Είχαμε μια συζήτηση μεταξύ μας, μεταξύ των δύο, σχετικά με τα, τις εναλλακτικέ ε, λύσεις. Ε, δηλαδή, μπορεί να έχουμε περισσότερο χρόνο αλλά ε, επιτόκιο ή ε, αντίστοιχα ναι να υπάρχει δυνατότητα για μικρότερο επιτόκιο αλλά τότε θα πρέπει να ε, είναι το χρονικό διάστημα πολύ πιο σύντομο. Άρα ή το ένα ή το άλλο και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Εμείς ως οι δύο οι συνεισηγητές ε, έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα ε, και ε, δεν θέλω να μπούμε σε τρομερές λεπτομέρειες γιατί θα ξαναρχίσουμε μεγάλη συζήτηση. Απλώς να σας πληροφορήσω ότι εμείς το συζητήσαμε το θέμα αυτό μεταξύ μας και είπαμε μία από τις δύο λύσεις. Ε, τώρα, ο κύριος Λούκα αναφέρθηκε στην ε, δομή της αγοράς, υπάρχουν όμως και άλλα ε, στοιχεία τα οποία ε, μπορούν να φέρουν ισορροπία ή όχι. Κοιτάξτε, ε, εάν, ε, εάν διαγραφεί αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα στην, στον κανονισμό και δουλέψουμε περισσότερο στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, κατά την άποψή μου θα ήταν πιο λογικό. Πάντως ε, νομίζω ότι όσον αφορά το περιεχόμενο, επί της ουσίας ε, έχουν ληφθεί υπόψη και συμπεριληφθεί οι ε, διάφορες συμβολές αυτά. Να ευχαριστήσω, κάτι που δεν έκανα την πρώτη φορά, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για όλη τη βοήθεια που μας έχουν δώσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ και εγώ με λίγο με αυτά που είπατε και τη λογική συσχέτιση μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους επιχειρηματολογίας σας γιατί το πρώτο είναι αυτό το, δημιουργεί το πρόβλημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε στο δεύτερο πέρα από τις διαφορές με τους Αμερικανούς αλλά αν θέλουμε να πιέσουμε την τράπεζα να κάνει hedge funding ε, αμέσως και μετά να προσφύγει σε έξι μήνες, τότε δεν είναι, θέλουν να πάρουν πίσω την εγγύηση, το, το, το ενέχειρο που έχει δοθεί και εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Και απ' την άλλη έχουμε ένα ε, σοβαρό σύστημα υποχρεωτικής κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αν ε, το συζητήσετε με τους εμπλεκομένους δεν είναι και τόσο μαλακό όσο λέτε εσείς γιατί και πάλι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ μέτρων πυλώνα 2 που είναι ανά άνοιγμα αναδάνειο και υπάρχει μια εποπτική προσδοκία που θα πει ότι ίσως να είναι καλό, ε, ε, δεν είναι ε, κόκκινο δάνειο γιατί καλύπτεται από καλό ενέχειρο. Όταν χρειάζεται ένα μέτρο υποχρεωτικό του πυλώνα 1, υποχρεωτικό για όλους, ανεξάρτητα από τα, την ιδιαιτερότητα του δανείου. Γι' αυτό και στο Συμβούλιο ε, είδαν πολύ θετικά το γεγονός ότι βρήκαμε μια λύση που ξεμπλοκάρει αυτούς τους φακέλους και πραγματικά με άνευ προηγουμένου ταχύτητα κινήθηκε και το Κοινοβούλιο και η Ένωση γενικά για να προσθέσει ένα στοιχείο στους τραπεζικούς κανόνες που πράγματι είναι ε, πολύ αποτελεσματικό. Κάνει διαφορά δηλαδή. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι πολύ επίοικες. Ήταν επώδυνος ο συμβιβασμός ίσως και για τις δύο πλευρές. Σίγουρα για την πλευρά μου. Και εξορισμού είναι, ε, ε, είναι ε, συμβιβασμός αυτός. Είναι κάτι που δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίοικης λύση. Αντίθετα μάλιστα. Είναι ισορροπημένη η λύση αυτή ε, βεβαίως εμείς ήρθαμε για να υπερασπιστούμε την πρότασή μας, θα διαβάσουμε και τις τροπολογίες σας βέβαια. Αλλά δείτε το με σοβαρότητα το θέμα, όχι ως ευκαιρία για προπαγάνδα, γιατί άμα κάνουμε προπαγάνδα, ο καθένας παίρνει τη θέση του και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα εγχείρημα άνευ προηγουμένου όπου σε λίγες εβδομάδες μόνο κάνουμε μεγάλη μεταρρύθμιση στους τραπεζικούς κανόνες και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Μπέρτ Λούκα. Το δίλημά σας είναι ακριβώς αυτό που αντιμετωπίζουμε. Από τη μία πλευρά δεν θέλουμε να δώσουμε ένα πλεονέκτημα στις μη ρυθμιζόμενες οντότητες που είπε όπως και η Γκουε είπε μπορεί να μην έχουν την καλύτερη διαχείριση του ενεχείρου γιατί θέλουν να πάρουν τα λεφτά και δεν τους νοιάζει αν πτωχεύσει η εταιρεία, άμα ε, δεν θέλουν πρόσθετη χρηματοδότηση γιατί, να δώσουν γιατί δεν είναι τράπεζες και ε, δεν θέλουμε βέβαια να δώσουμε χώρο για καταστρατήγηση όπου θα αρχίσουν να ε, πασάρουν η μία τράπεζα στην άλλη το δάνειο. Πρέπει να βρεθεί μια σοβαρή λύση. Πιστεύω λοιπόν ότι Α, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη στο κείμενο του Συμβουλίου που είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Εμεί το έχουμε βάλει όπως είναι και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ένα πράγμα είναι αν το ημερολογιακό έτος αρχίζει από το έτο 1, αλλά αρχίζει, ε, λαμβάνει υπόψη όμως την ε, ε, απαξίωση του δανείου Οπότε αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά αφήνει λίγο ανοιχτά το πρόβλημα για τα μη ε, ασφαλισμένα ε, ανοίγματα. Εκεί έχουμε ένα περιθώριο ελιγμών που την προβλέπει η, το που το προβλέπει η καμπύλη μας. Ε, θέλουμε, έτσι μπορούμε να έχουμε ίσους κανόνες του παιχνιδιού και να αποφύγουμε παραθυράκια καταστρατήγησης των κανόνων αυτό θα το επεξεργαστούμε περισσότερο και είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και σε επικοδομητικές σκέψεις από την πλευρά σας για να βρεθεί μια λύση γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επί του στόχου και επί των διασφαλίσεων αλλά πρέπει να βρεθεί η σωστή λύση. Το Συμβούλιο δεν βρήκε γιατί δεν είναι εύκολη η εξέβρεση λύσης ε, αλλά θα ήταν καλή συνεισφορά του Κοινοβουλίου αν μπορούσαμε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση στο ζήτημα αυτό και βέβαια θα δούμε όλες τις τροπολογίες και τα πρόσθετα στοιχεία της κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση για την κοινωνική ασφάλιση γιατί εδώ είναι ένας προληπτικός κανονισμός, ε, πρέπει να ετοιμαστεί και η οδηγία για να ενισχύσουμε τη λογική μας. Ευχαριστώ πολύ. Η 23 Νοεμβρίου η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στις 12 και Καλό είναι να είναι στα αγγλικά οι τροπολογίες για να μας διευκολύνεται. Οπότε στις 6 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα διάλειμμα μέχρι στις 2.30 με δημόσια κρόαση με την Ντανιέλ Νουή και μετά στις 4 έχουμε τον Ανδρέα Ενρία για το, τη διαδικασία του διορισμού. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε.